Ε, μία νέα διάταξη, ασυνήθι θα έλεγα. Ελπίζω να υπάρχει επαρκής χώρος. Σε αυτή την τελευταία μας συνεδρία, σε πριν από τα Χριστούγεννα. Ε, ησυχία παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε, ελπίζω ναι. Ε, χρειάζομαι κι άλλη για να δω τον Κυριάκο που κάθεται εκεί απέναντι. Η τελευταία φορά που ήρθαμε στην αίθουσα αυτή είχαμε την συνάντηση, τη διάσκεψη με την Επιτροπή και τη διάσκεψη των Προέδρων και όλη η Κομισιόν καθόταν από αυτή την πλευρά και εμείς από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλωσορίζω όλους πολύ θερμά στην τελευταία μας συνεδρίαση του 2011 που νομίζω ότι ήταν ένα έτος πετυχημένο θα έλεγα και με μεγάλη δραστηριότητα για την Επιτροπή μας η Πολωνική Προεδρία στήριξε το έργο μας της εσωτερικής αγοράς και το, όχι μόνο με το φόρουμ που οργανώθηκε στην Κρακοβία για την εσωτερική αγορά, αλλά γενικότερα. Και νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε την Πολωνική Προεδρία για το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πράξης για την ενιαία αγορά είναι το πρώτο θέμα της ατζέντα για την ανάπτυξη. Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από, το και από τους υπουργούς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μας στον αναπληρωτή πρωθυπουργό, τον κύριο Πάμπλακ, ο οποίος ήρθε στη συνεδρίασή μας, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους σας που συνέβαλαν. Αυτά ως μια σύντομη εισαγωγή. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερησιά διάταξη, εντάξει, και να σας πω ότι η συνεδρίαση αυτή εκπέμπεται μέσω του διαδικτύου. Ελπίζω οι συνάδελφοι να μας παρακολουθούν online και να μην έχουν πάει έξω για χριστουγεννιάτικα ψώνια. Καταρχήν θα ακούσουμε την παρουσίαση του συμπερασμάτου της Πολωνικής Προεδρίας και θα είναι εδώ ο Γκρέκ, ο κύριος Ρο Κούχολα. είναι σε μια επιτροπή, η κυρία είναι στην Επιτροπή Βιομηχανίας για, σε μια συνεδρίαση που ασχολούται ασχολείται με την περιαγωγή και η κυρία Βανίρ στη συνέχεια ε, θα ε, ασχοληθεί με την ανακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών για την τροποποίηση του κανονισμού, μετά τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά. Ε, η κυρία Ιβανόβα και μετά όπως είπα περιαγωγή από την κυρία Κόρχολα. Και σήμερα το απόγευμα, τέλος, θα πιούμε ένα ποτήρι μαζί στις 6.30 έξω από την αίθουσά μας. Όχι μόνο για να γιορτάσουμε ένα πετυχημένο έτος, αλλά και επειδή ε, ως επικεφαλής ε, της ε, Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ο Herbert Γέννητ θα είναι μαζί μας. Πράγματι, ε, ήταν πολύτιμη η συμβολή και η συνεισφορά του ε, στο έργο της ε, ΙΜΚΟ. Και παρακαλούμε και όλους τους φίλους και τους ενδιαφερόμενους να έρθουν μαζί μας να πιούν ένα ποτήρι κρασί στις 30 όπως είπα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγικά και αμέσως τώρα καλωσορίζω την κυρία Αντόσκα και την κυρία Τόμκιλ η κυρία Τόμ Κιλ έχει έρθει και προηγουμένως με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό. Με την κυρία Κρασνότσκα έχουμε συνεργαστεί ε, και τώρα δίνω αμέσω το λόγο στην κυρία Χεν Κλιόσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τιμή και ευχαρίστηση να σας απευθύνω το λόγο εξ ονόματος της πολωνικής ε, κυβέρνησης και να μιλήσω για τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Πολωνικής Προεδρίας σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Ελπίζω ότι όλες οι προσπάθειες που καταβάλαμε για να ενισχύσουμε την συνοχή της κοινής εσωτερικής αγοράς θα ε, προσφέρουν απτά θετικά αποτελέσματα και στις εταιρείες αλλά και στους πολίτες και τους καταναλωτές. Εμείς δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εσωτερική αγορά, γι' αυτό και δρομολογήσαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως κινητήριος δύναμης για την ανάπτυξη. Η ενιαία αγορά πάντοτε υπήρξε στο επίκεντρο της προσοχής μας. Έπρεπε να λειτουργήσουμε βέβαια υπό δυσμενέστατες συνθήκες. Φέτος τον Ιούλιο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο κύριος Παύλακ, παρουσίασε το νοδικό μας χάρτη, το πρόγραμμά μας της Πολωνικής Προεδρίας. Μετά, τον Ιούλιο βέβαια, κανένας δεν ανέμενε ότι η Ευρωζώνη θα βρεθεί σε μία περίοδο αναταραχής. Οι χρηματοοικονομικές αγορές παρατηρούσαν από πολύ κοντά το τι ακριβώς συνέβαινε κατά τις διαδοχικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έτσι η Πολωνική Προεδρία έπρεπε να εστιάσει όλη της την προσοχή στο να ενισχύσει την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι μια ισχυρή εσωτερική αγορά θα διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Είναι ε, καθοριστικής να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης και είναι υψίστης σημασία να ε, δώσουμε νέα όθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την έρευνα ετήσιας ανάπτυξης που πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα αυτή συστήνει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους τομείς που βαίνουν προς την ανάπτυξη, να καταργήσουμε όλα τα εμπόδια, να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πατέντα, να ε, εφαρμόσουμε την οδηγία των υπηρεσιών και να οθήσουμε την ψηφιακή κοινή αγορά. Δηλαδή, να βρούμε ε, συμβιβαστικές λύσεις στις πρωτοβουλίες εκείνες οι οποίες θα ενισχύσουν την οικονομική μας ανάπτυξη το ταχύτερο δυνατό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Πολωνική Προεδρία αναζήτησε την ε, ταχύτερη, γοργότερη εφαρμογή όλων των πρωτοβουλειών της ε, πράξης της ενιαίας αγοράς. Και με ικανοποίηση μπορώ να αναφέρω ότι η Πολωνική Προεδρία ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο σε ένα βασικό θέμα. Και αυτή είναι η ενιαία ευρωπαϊκή πατέντα. Λοιπόν, αναφερόμαστε στο ενιαίο ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό δίπλωμα Ξέρω ότι ε, όλα αυτά δεν ανήκουν ε, ακριβώς στην αρμοδιότητά σας. Απλώς θέλω να πω ότι η συμφωνία που επιτεύθηκε ε, θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους κατά 80%. Τούτο σημαίνει ότι οι εταιρείε μας θα έχουν ένα, στη διάθεσή τους ένα σύστημα, ένα σύστημα ενιαίο ε, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύστημα ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτό έγινε και με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έτσι δίδεται και η ιδιαίτερη ευκολία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Καταβάλαμε επίσης τεράστια προσπάθεια σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες ε, ε, για την επίλυση της διαφοράς επί των διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έξι μήνες διήρκησε η όλη προσπάθεια και τελικά κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση σε όλα τα θεμελιώδη ζητήματα. Το μόνο θέμα το οποίο ακόμα εκκρεμεί είναι η έδρα αυτού του δικαστηρίου ε, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Τεχνίας. Μετά από 8 ε, χρόνια λοιπόν διαπραγματεύσεων καταλήξαμε. Υπάρχει και μια άλλη προτεραιότητα της ε, πράξης της ενίας αγοράς. Αφορά την τυποποίηση και τον σχετικό ε, κανονισμό ε, με την τυποποίηση. Άρχισαν λοιπόν οι διαπραγματεύσει, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ώστε να επιτευχθεί η τελική συμβιβαστική λύση κατά την πρώτη ανάγνωση υπό την Δανέζικη Προεδρία. Ε, περιμένουμε να δούμε τι θα υποβάλει η κυρία Λάρα ακόμη. Η έκθεση θα είναι στη διάθεσή μας τον Ιανουάριο του 12. Έχει σημειωθεί επίσης σημαντική πρόοδος σε ένα σχέδιο κανονισμού που αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εσωτερική αγορά. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συνεργασία μεταξύ Δανέζικης Προεδρίας και του εισηγητή κυρίου Άνταμ Μπιελάν θα καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία θα επιτευχθεί κατά το πρώτο εξάμεινο του προσεχούς έτους. Επίσης, συνεχίσαμε το έργο και τη δραστηριότητά μας σε διάφορα θέματα τεχνικής φύσεως, τεχνικής νομοθεσίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλβατόρε Ταταρέλα. Οφείλουμε στη δική του αποφασιστικότητα το γεγονός ότι η Πολωνική Προεδρία συνέβαλε στην ε, ε, έκδοση ε, ενός σχεδίου οδηγίας σχετικά με τα καυσαέρια των μικρού μεγέθους γεωργικών μηχανημάτων. Ε, στο Συμβούλιο τώρα. Είχαμε στενή συνεργασία με τον κύριο Παντζέρη, τον εισηγητή και συνεργαστήκαμε ε, και σε σχέση με το κανονισμό σχετικά με τα οχήματα τα δύο, τριών και τεσσάρων τροχών. Η Πολωνική Προεδρία ξεκίνησε επίσης δρομολόγησε το σχέδιο οδηγίας ε, σχετικά με τα σκάφη αναψυχής και τα σκούτερς ε, θαλάσσης. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Χάρμπορ και σίγουρα θα συνεργαστούμε και με την Δανέζικη Προεδρία. Και ξεκινήσαμε επίσης και τις διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την περιαγωγή, το roaming. Ε, αναμενόταν πάρα πολύ αυτή η πρόοδος και η Πολωνική Προεδρία ε, λίανε αν θέλετε το δρόμο για την Δανέζικη Προεδρία ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία πριν εκπνεύσει η αρχική οδηγία τον Ιούνιο του 12. Εκτιμούμε λοιπόν όλες τις προσπάθειες της κυρίας Κορχόλα, η οποία υπήρξε εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Την ευχαριστούμε θερμά. Η Πορωνική Προεδρία κατέβαλε επίσης ε, μεγάλη προσπάθεια στο ε, θέμα της εφαρμογής των πνευματικών δικαιωμάτων στα τελωνία των κανονισμών των σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, οργανώσαμε και μία δημόσια ακρόαση στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό διότι ε, αποδείχθηκε σε ποια πράγματα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ας πούμε, ε, σε θέματα παράλληλων αναθέσεων κλπ. Επίσης, είχαμε μια συζήτηση τρογγυλής του τραπέζης υπό την προεδρία του κυρίου Κλόιτσμαν και την κυρία Μάριν Γκαγιό. Αναλήφθησαν και άλλες πρωτοβουλίες που συνέπεσαν με τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή, με τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχει το θέμα των νέων οδηγιών που θα πρέπει να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς για το μάρκετινγκ προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνική Προεδρία ξεκίνησε επίσης να δουλεύει σε ολόκληρο το πακέτο. Συζητούμε τα βασικά θέματα, αλλά όχι τις οδηγίες αυτές καθευτές. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει, προσεγγίζει το πακέτο στο σύνολό του. Ε, πιστεύουμε ότι διευκολύναμε αρκετά το έργο αυτών που θα ακολουθήσουν. Επίσης, το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής και το σχετικό ε, νομικό πλαίσιο είναι ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε. Θέλουμε να υπάρξει εναρμόνιση, γι' αυτό οργανώσαμε ένα συνέδριο στις 9 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία, όπου ακριβώς συζητήθηκε το θέμα αυτό. Αναμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον είδαμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Κατά τη γνώμη της Πολωνικής Προεδρίας, η ανάλυση της εμπειρίας που συσσωλεύσαμε σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάλυση αυτή είναι πολύ σημαντική και πολύ απαραίτητη. Απαιτούνται δράσεις που θα βελτιώσουν την κινητικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα στα επαγγέλματα που είναι ρυθμισμένα. Η Πολωνική Προεδρία βεβαίως δεν μπορούσε να κάνει τα πάντα. Υπήρξαν καθυστερήσεις στις, στην έκδοση ανακοινώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν και δεν ξεκινήσαμε, δεν δρομολογήσαμε τη συζήτηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο ελπίζουμε ότι η Δανέζικη Προεδρία η οποία ακολουθεί θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Και αξίζει να σημειωθεί νομίζω ότι οι πάντες στην εσωτερική αγορά ενδιαφέρονται για τη συζήτηση αυτή και για τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δηλαδή αυτό των καθυστερήσεων, δεν μπορέσαμε να ξεκινήσουμε το έργο σε άλλους τομείς προτεραιότητες, όπως είναι οι κρατικές προμήθειες. Συνοπτικά, κυρίες και κύριοι, και εν κατακλείδη θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για ένα γεγονός που συζητήθηκε ευρέως αυτή την Επιτροπή. Τόσο η Πολωνική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η ΙΜΚΟ, μπορούν να είναι υπερήφανοι, διότι οργανώσαμε το πρώτο φόρουμ ενιαίας αγοράς. Οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πολωνική Προεδρία. Πρόκειτο για μια κοινή προσπάθεια από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε την εκδήλωση αυτή στην Κρακοβία. Πάνω από 1.200 συμμετέχοντες συνέβαλαν, συμμετείχαν στη συζήτηση για την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς. Εκπρόσωποι εργοδοτών, ε, εργατικών σωματείων, επιμελητηρίων, εμπορικών και άλλων, ε, επιστήμονες, επιχειρηματίες. Είχαμε δηλαδή μια πολύ πλούσια εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ και επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ρουζατούν και όλους όσοι στην Επιτροπή ΙΜΚΟ μας βοήθησαν στη διοργάνωση που μας στήριξαν ανεπιφύλακτα καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της εκδήλωσης. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 1η ε, Δεκεμβρίου σχετικά με τα αποτελέσματα του φόρουμ. Και η διακήρυξη η οποία θετήθηκε στο τέλος του φόρουμ συγκέντρωσε την υποστήριξη όλων των κρατών μελών. Η Πολωνική Προεδρία δεν το περιέλαβε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό το Συμβούλιο συνήλθε στις 5 Δεκεμβρίου και με ικανοποίηση εγκρίθηκε και η διακήρυξη της Κρακοβίας εγκρίθηκε μάλλον το περιεχόμενο της διακήρυξης και αποφασίστηκε να υπάρξει και ένα follow-up, μια συνέχεια του χρόνου. Ε, η 20η επέτειος θα γιορταστεί της ε, εσωτερικής αγοράς του χρόνου. Ε, τέλος, εξασφαλίστηκε η δέσμευση των χωρών μελών για την κατάργηση εξάλληψη όλων των σοβαρών ε, προσκομμάτων και φραγμών που ισχύουν, υπάρχουν ακόμα στην εσωτερική αγορά. Ε, στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου νομίζω ότι αναδείχθηκε μια νέα διάσταση, μια διάσταση ποιότητας, γιατί δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουν αυτοί για τους οποίους ε, ουσιαστικά δημιουργήθηκε αυτός ο νέος κανονισμός. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι τα όσα σας ανέφερα, τα επιτέγματα της Πολωνικής Προεδρίας αποδεικνύουν επαρκώς ότι η ενιαία αγορά υπήρξε πράγματι τομέας προτεραιότητας για την Προεδρία μας, για την Πολωνική Προεδρία προσπαθήσαμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό, ώστε η ευρωπαϊκή αγορά να γίνει πιο προσβάσιμη, προσπελάσιμη προς τις εταιρείες και τους πολίτες μας. Ελπίζω ότι οι επόμενες προεδρίες, οι Δανέζικοι και στη συνέχεια η Κυπριακοί ασφαλώς θα χρησιμοποιήσουν τους καρπούς και τα αποτελέσματα του έργου μας και θα φέρουν αυτή την προσπάθεια σε νέα φάση. Ευχαριστώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξαιρετική συνεργασία με την Προεδρία αλλά και με όλους τους εμπειρογνώμονες. Με ικανοποίηση αντιλαμβάνομαι ότι είστε σύμμαχοί μας υπέρ της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Τώρα, εάν νομίζετε ότι δεν αναφέρθηκα επαρκώς σε κάποια από τα θέματα που απασχολούν την ενιαία εσωτερική αγορά. Είμαι έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Really, my introduction when I said what a strong supporter of the single market the presidency had been, and I think if I particularly mention the single market forum, I think we were very pleased to see the resolution there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 απασχόλησαν και τους καταναλωτές και τη συμπεριφορά τους στην αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι μηχανισμούς έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεμονωμένες απειλές. Γιατί πιστεύω ότι οι καταναλωτές αν έχουν τα κατάλληλα μέσα μπορούν να συνεισφέρουν και στην οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό η Πολωνική Προεδρία μπορεί να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, να προωθήσει την ασφάλεια και την προστασία. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας, δηλαδή η περαιτέρω εξέταση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, διότι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και με τις δραστηριότητες αυτές ε, θέλαμε να απευθυνθούμε στον ε, να προασπίσουμε μάλλον την αρχή της ενιαίας αγοράς όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταναλωτές. της 11 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Θέλουμε λοιπόν να επικεντρώσουμε την προσοχή στους καταναλωτές που θα έχουν ρόλο ζωτική σημασία στην ενιαία αγορά. Γι' αυτό ως Προεδρία υποστηρίξαμε τις εργασίες αυτές, οργανώσαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έλαβε χώρα στην ομάδα εργασίας υπέρ των καταναλωτών και πληροφόρησή τους στις 21 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα τεχνικής υφής έγγραφο για τις δραστηριότητες που προβλέπονται. Στην ομάδα εργασίας υποστηρίχθηκε το πρόγραμμα αυτό και μιλήσαμε και για την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στους διάφορους τομείς. Θα υποστηρίξουμε βεβαίως και την Προεδρία της Δανίας κατά το προσέχες εξάμεινο. Επίσης, μας απασχόλησε η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η αποδοχή της έγινε στις 10 Οκτωβρίου, στις 22 Νοεμβρίου. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη-μέλη έχουν χρόνο μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου του 2013 για να εντάξουν την οδηγία στην εσωτερική ένωμη τάξη τους. Όπως γνωρίζετε, οι τριετής αυτές διαπραγματεύσεις ήταν δυσχερείς, προβλέφθησαν πολλές δράσεις και πολλές φορές είχαμε διφορούμενες αποφάσεις. Η ΙΜΚΟ υπό τον Μάλκομ Χάρμπορ επιτέλεσε ένα πολύ θετικό έργο. Και το ίδιο αφορά και τον Ανδρέα Σβάμπ και τους Σκιώδης. Έτσι μιλάμε για μία εξισορρόπηση της προστασίας των καταναλωτών και των ενιαίων ρυθμιστικών πλαισίων υπέρ αυτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προκατόχους, ιδιαίτερα την Ουγγρική Προεδρία. Ελπίζουμε αυτό το μέσο να δώσει μία όθηση στην αγορά και να δώσει εγγυήσει στους καταναλωτές για μια σχετική άνεση. Επίσης, ελπίζουμε να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές συναλλαγές. Με βάση αυτή την πρόκληση και για να την αντιμετωπίσουμε, προβλέπουμε ένα πρόγραμμα έτσι ώστε οι καταναλωτές να επιλύουν τις διαφορές τους. Αυτό αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας μέσα στα πλαίσια του, της πράξης ενιαίας αγοράς. Και υπάρχει και η απόφαση της Κομισιόν για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών ή τις επιγραμμικές, την επιγραμμική επίλυση διαφορών. Μιλήσαμε για τα σεμινάρια αυτά που οργανώθηκαν στην Κρακοβία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ροζατούν για την πρωτοβουλία της και για το έργο της γενικότερα. Στη συνέχεια συντάχθηκε και η δήλωση της Κρακοβίας, όπου μιλάμε για προτεραιότητες, για... Μιλάμε για πρωτοβουλίες για την επίλυση διαφορών. είτε γίνεται online είτε στην αλόδαπη. Επίσης, μιλάμε για τα εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την διαφοροποίηση στις ε, επιμερούς χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, ένα ευρύ ποιοτικό φάσμα. Ποιοτικά κριτήρια δηλαδή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να κατανοηθεί το θέμα επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών, πολιτών δηλαδή και επιχειρήσεων Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αγορά συμμετέχουν στο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτό το σύστημα επίλυσης διαφορών επιγραμμικά έτσι ώστε να βοηθήσουμε και στην ενιαία, στη συγκρότηση της ενιαίας ηλεκτρονικής αγοράς τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στο νομοθετικό πακέτο που παρουσιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών ή την επίλυση διαφορών online επιγραμμικά. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 5 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκαν αυτά τα δεδομένα. Η την επιλυση διαφορων online επιγραμμικα στο συμβουλιο Ανταγωνιστικό σας 5 Προεδρία θα ήθελε να συζητήσουμε καταρχήν τις προτάσεις της Κομισιόν. Αυτό έγινε στις ομάδες εργασίας ε, στη... για την προστασία του καταναλωτή και στις 29 Νοεμβρίου παρουσιάσαμε αυτά τα σχέδια. Έτσι, τα κράτη-μέλη εκφράστηκαν αρχικά στις 13 και 14 Δεκεμβρίου. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις και έγινε η πρώτη συζήτηση για το πακέτο στο σύνολό του, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό. Μιλήσαμε για ένα συμβασμό μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών και δίνουμε και τα πρώτα αποτελέσματα προς την Δανέζικη Προεδρία για αυτό το νομοθετικό κείμενο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια τελική μορφή του κειμένου, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Σας εύχομαι ε, καλή ε, συνεργασία και αποτελέσματα. Αυτά προς την κυρία Ρόζα Τούν και τον κύριο Γκρέγκ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ε, επιλύσουμε τις διαφορές επιγραμμικά, κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα επικοδημητικό για τους καταναλωτές και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη, για τις προσεχείς προεδρίες. Ως υπεύθυνη για την προστασία των καταναλωτών, κατά την Πολωνική Προεδρία, ορίσαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα για την ανταγωνιστικότητα και τους καταναλωτές, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Χωακίν Αλμούνια ήταν υπεύθυνος από πλευράς ε, Κομισιόν και ο Ανδρέας Σβάμπ από πλευράς ε, εισηγητών από το Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια ελεύθερη αγορά και για μηχανισμούς που βρίσκονται στα χέρια των καταναλωτών. Όπως είπε και ο κύριος Σβάμπ, οι στόχοι της ε, μακροχρόνιας πολιτικής ανταγωνισμού ε, αποτελούν ευεργέτημα για όλους τους συμμετέχοντες. Μιλάμε για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, γιατί αντίθετα θα ήταν κάτι το επιζήμιο και για τους καταναλωτές και για την οικονομία. Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική προστασία των καταναλωτών μπορεί να βοηθήσει στην ποιότητα ζωής των ε, καταναλωτών. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί. με βάση και τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Να έχουμε δηλαδή μία ευφυή ανάπτυξη και μία ισορροπημένη ανάπτυξη για την κοινωνία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καταναλωτές που την χάνουν προστασίας και που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό θα θέλαμε να ενισχύσουμε τη θέση τους και να τους προσφέρουμε όλα τα, τα σχετικά θετικά στοιχεία και ευεργετήματα. Αυτό θα γίνει κατά τα προσεχή έτη και ελπίζω η αναθεώρηση των ε, διαφόρων οδηγιών να βοηθήσει τους καταναλωτές και μέσα στα πλαίσια του 2014-2020. Ελπίζω να έχουμε αίσιο πέρας και ελπίζω να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα στα πλαίσια αυτής της Τρόικας, των τριών προεδριών δηλαδή. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας. Τέλος, θα ήθελα να, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για το προσεχές έτος. Ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ και τις δυο σας και για τα όσα μας είπατε και για τις ευχές σας και για το υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο που μας υπενθυμίζει τα πολωνικά Χριστούγεννα και είναι εκτός του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αρχίσατε να προχωράτε τις νέες προτάσεις και έχετε και μια παρουσίαση για την αξιολόγηση που και πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο είναι ελαφρώ πιο μπροστά από το Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Ελπίζω να δώσετε λοιπόν το καλό παράδειγμα στη Ιδανική Προεδρία. Θα κάνουμε και εμείς παρουσίαση της αξιολόγησης αντικτύπου με τους δύο εισηγητές, ε, τον κύριο Γκρέχ και την κυρία Τούρν που είναι εδώ. Και να πω για το φόρουμ η συνεισφορά σας όπως και της κυρίας Τούρ και του κυρίου Γκρέχ αλλά και όλων όσων ε, είναι εδώ ε, ήταν που και ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Είναι πολύ σημαντική. Είχαμε μια πολύ σημαντική παρουσίαση των 20 ε, βασικών ανησυχιών των πολιτών στην νέα αγορά, κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και είναι κάτι το οποίο έλειπε από το Φόρουμ της Ενιαίας Αγοράς. Θα δώσω τώρα το λόγο για ερωτήσεις και σχόλια από την Επιτροπή. Έχουμε τους ε, συντονιστέ μας, τον κύριο Σφάμπ, την κυρία Γκέμπχαρτ, τον κύριο Κρόιτσμαν. Θέλει να λάβει το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σβάμπ. Μετά η κυρία Γκέπχαρτ και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ πολύ, κυρίες μου. Έχω δύο ε, πολύ σύντομα σχόλια να κάνω. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας ε, στη διάρκεια του προηγουμένου εξαμήνου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος του ΕΛΚΘΕ. Η Πολωνία, η πολωνική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι είχαν προεκλογική εκστρατεία και εκλογές, ε, προσέδωσαν μεγάλη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Υπάρχουν τρία ε, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αναφερθήκατε στο φόρουμ της εσωτερικής αγοράς. Ε, αυτό που είπε η Υπουργό ελπίζω να επαληθευτεί. Ελπίζω δηλαδή να έχουμε τον κανονισμό στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ομοιομορφία στου κανόνε τη εσωτερική αγορά. Ελπίζω να συνεχίσετε να προασπίζετε τα θέματα αυτά με ενεργό τρόπο στο Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος είπε άλλωστε ότι ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμβαδίζουν για τα θέματα αυτά και αν συμβαδίζουν μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα την ε, ε, συνεργασία και την αρμόδια αρχή για την προστασία των καταναλωτών, η ισορροπία σε θέματα ανταγωνισμού και καταναλωτών είναι πολύ σημαντικά. Η εκδήλωση του να με εντυπωσίασε γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορούν τους, πολι... τους καταναλωτές είτε άμεσα είτε έμεσα, ε, αλλά πολλές φορές όλα αυτά είναι κατακαιρματισμένα σε διαφορετικά τμήματα. Αν καταφέρουμε να έχουμε μια οριζόντια πολιτική θα ήταν κάτι πολύ επιτυχές, όπως κάνατε στην Πολωνία. Ε, και αυτό θα ήταν καλό και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Η συζήτηση δε για την οδηγία για τις υπηρεσίες, όπως είπε και η κυρία Χάνσλικ στην έκθεσή της, ήταν πολύ σημαντική, όπως και η συζήτηση για τις ε, υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα ενίας αγοράς είναι πολύ σημαντικά και σχετίζονται με την ε, Προεδρία σας. Ε, θέλουμε να αναγνωριστούν άλλωστε τα επαγγελματικά προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμεθοριακά και θέλουμε να έχουμε μια αγορά απασχόλησης, μια εσωτερική αγορά απασχόλησης. Ελπίζω οι Δανείοι να αναλάβουν τα ενία από εκεί που έχετε σταματήσει και προσβλέπω ε, στη συνεργασία με τη νέα Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις εκπροσώπους ε, της Πολωνικής Προεδρίας. Ε, χαίρομαι πάντα όταν ε, έχουμε γυναίκες ανάμεσά μας, διότι σε επίπεδο κυβερνήσεων στην ευρωπαϊκή πολιτική δυστυχώς πολύ συχνά κυριαρχεί η ανδρική παρουσία. Γι' αυτό λοιπόν με χαροποιεί ιδιαίτερα όταν είναι τόσο ε, καλές ε, στο καθήκοντα αυτά γυναίκες. Ε, χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για αυτό το γεγονό. Βεβαίως υπήρχαν και άνδρες εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης, με πρώτο τον κύριο Τάσκ, Τούσκ. Ε, πρόκειται για μια προεδρία βέβαια που επικεντρώθηκε πολύ στις ευρωπαϊκές πτυχές και ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι, είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις να υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μας μας δόθηκε η αίσθηση ότι με αυτή την Προεδρία και με τον ε, συγκεκριμένο Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό ακριβώς ε, συνέβη. Ελπίζω να αποτελεί αυτό ευίωνο μήνυμα για το μέλλον και ελπίζω και οι μελλοντικέ ε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κάνουν εξίσου πολλά πράγματα με την Πολωνική Προεδρία. Δυστυχώ πάντα δεν συνέβαινε αυτό. Είχαμε το φόρουμ για την ενιαία αγορά και ήταν το πρώτο φόρουμ αυτή τη μορφή. Και προέκυψε κάτι το οποίο ε, συνήθως δεν κάνουμε ποτέ. Βάλαμε στο επίκεντρο τον καταναλωτή. Με αυτά τα 20 αιτήματα των πολιτών καταφέραμε να αποδείξουμε πού ε, έγινε τα προβλήματα. Και αυτό φυσικά μας απέδειξε ότι οι πολίτες θέλουν περισσότερη Ευρώπη και επιθυμούν να κινηθούν προς μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιη ότι η Δανέζικη Προεδρία θα αναλάβει ε, τα ενία από εκεί που ε, σταμάτησε η Πολωνική Προεδρία και θα συνεχίσει με όλες τις προκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί την επόμενη χρονιά. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι η προστασία των καταναλωτών. Μόλις αναφερθήκατε σε αυτό και εσείς, η προστασία των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική ώστε οι πολίτες να εμπιστεύονται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εμπιστεύονται ε, τις αγορές ε, σε άλλες χώρες. Να μπορούν λοιπόν να δραστηριοποιούνται ως καταναλωτές και διαμεθοριακά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ως αντιπροσωπεία μιλούσαμε με οργανώσεις καταναλωτών, ε, διαπίστωσα και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για σας, ότι πρέπει να εργαστούμε πολύ περισσότερο και να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο με τις οργανώσεις καταναλωτές καταναλωτών, ώστε να βρούμε τι κατάλληλε απαντήσει. Και αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε προ αυτή την κατεύθυνση και στην Πολωνία και σε άλλε χώρε, σίγουρα θα προκύψει κάτι πολύ θετικό. Και νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το εξάμεινο, το οποίο πράγματι υπήρξε πολύ παραγωγικό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Κρότσμαν και στη συνέχεια η κυρία Τούτ. κάποιο άλλο θέλει να λάβει το λόγο, ο κύριο Κρότσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία για την αφοσίωση και δέσμευση που επέδειξε και στη Ρόκλαο και στην Κρακοβία και στη Βαρσοβία το διαπίστωσα αυτό. Ε, είναι παράδειγμα το οποίο μπορούν να ακολουθήσουν και οι άλλες χώρες μέλη. Ε, ξεπλάγει ευχάριστα στη Βαρσοβία όταν είδα πώς ε, δούλευαν όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό και είναι πράγματι, ήταν πράγματι πολύ εντυπωσιακό. Ε, τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι η προσπάθεια που κατέβαλε η Πολωνία υπέρ της Ευρώπης πραγματικά κατέπληξε όλους και ελπίζω να αποτελέσει παράδειγμα για τις άλλες προεδρίες. Ευχαριστώ η κυρία Τιούν και μετά η κυρία Βανιούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ δράτω με τις ευκαιρίες αυτής για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου όχι μόνο για τα ευγενικά λόγια αλλά εγώ συμμετείχα σε εκδηλώσεις ε, αυτής της ε, Προεδρίας. Πήγαμε και μία, ε, κάναμε και μία επίσκεψη μελέτη στην Κρακοβία και την Βαρσοβία και είναι πολύ ευχάριστη η ανάμνηση από τους συναδέλφους που συνάντησα αλλά και από τις συναντήσεις που είχα μαζί σας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν που ήταν τόσο δραστήριοι και ελπίζω ότι αυτή την ανταλλαγή θα τη συνεχίσουμε. Ιδιαίτερα στην Κρακοβία συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους και ελπίζω να τους ξανασυναντήσω. Και τα στελέχη, το προσωπικό, και δεν το αναφέραμε αυτό, πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή η προσπάθεια που κατέβαλαν. Πολλοί κόσμος πήγε στο φόρουμ στην Κρακοβία. Αυτό απαιτούσε τεράστια οργάνωση από το προσωπικό και με την ευκαιρία αυτή εκφράζω τις ευχαριστίες μου γιατί μέχρι τώρα δεν το κάναμε αυτό. Ελπίζω όπως είπα δεν είμαι πολύ αντικειμενική αλλά είδα αυτή την απίστευση, απίστευτη συγγνώμη, εμπλοκή της Πολωνικής Προεδρίας υπέρ της Ευρώπης, όπως επεσήμανε η κυρία Γκέπχαρτ. Η ευρωπαϊκή διάσταση, η, η διάσταση της αλληλεγγύης. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί με τις ε, προεδρίες που διαδέχονται την Πολωνική. Ενώ και το φόρουμ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ θετική εμπειρία και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε αυτά τα φόρα. Διότι τούτο είναι το πιο σημαντικό για την ενιαία αγορά μας. Δηλαδή να εμπλέκονται οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, η διοίκηση και η οργάνωση ενός τέτοιου φόρουμ ήταν πολύ χρήσιμη. Εγώ το στηρίζω για ένα, ως ένα project που πρέπει να συνεχιστεί και που θα δώσει αποτελέσματα. Ελπίζω να το συνεχίσουμε μία φορά το χρόνο ή κάθε δύο χρόνια ή όπως αλλιώς αποφασίσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κτίζουμε πάνω σε αυτό το οποίο ήδη επιτύχαμε. Να έχουμε ένα καλύτερο φόρουμ το 12 και ένα ακόμα καλύτερο το 13 κλπ. Με την ευκαιρία αυτή σας εύχομαι όλους καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό είναι να το οργανώνουμε κάθε δύο χρόνια. Η κυρία Βανιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά την Πολωνική Προεδρία. Εγώ είμαι Γαλλίδα και νομίζω ότι διδαχθήκαμε πολλά από την Προεδρία σας, διότι η Γαλλία βεβαίως είναι ιδρυτικό μέλος, αλλά μερικές φορές οι Γάλλοι πολίτες είναι τα κακομαθημένα παιδιά της Ευρώπης και ε, καμιά φορά ξεχνάμε το τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι ή σε τι Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνατε για την ενιαία αγορά. Διδάξατε και καθορίσατε ή μάλλον χαράξατε ξεκάθαρες ε, γραμμές ε, συνεργαστήκαμε αρμονικά με ένα πνεύμα συνεργασίας. Σας ευχαριστώ προσωπικά για το γεγονός ότι δόθηκε όθηση και λύθηκε το ζήτημα των διπλωμάτων ευρεστιχνέας, διότι σε περιόδους κρίσης ακριβώς αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, η ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Εγώ τώρα είμαι η συγγήτρια για την αναγνώριση των προσόντων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αγορά και για την ανάπτυξη αλλά και το δικαίωμα των εργαζομένων. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας διότι η οδηγία εκδόθηκε χθες αλλά βεβαίως και η Δανέζικη Προεδρία Υιοθετώντας τις προτεραιότητες αυτές θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε η Ανατολή με τη Δύση. Εσείς ανοίξατε το δρόμο και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Ρόιτερ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να προσθέσω λίγα λόγια προς την Πολωνική Προεδρία. Όλοι αναμέναμε ότι μια μεγάλη χώρα όπως η, η Πολωνία θα χρησιμοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για την επιτυχή έκβαση της Πολωνικής Προεδρίας. Πράγματι αυτό συνέβη. Όπως επίσης και οι Πολωνοί βουλευτές ε, εκπροσώπησαν την Πολωνία ως μια χώρα ενωμένη η οποία γνωρίζει προς τα που κατευθύνεται και θα ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ γι' αυτό. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας, τα οποία συμμερίζομαι και εγώ. Όπως βλέπετε, προχωρήσαμε πολλούς φακέλους και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό. Με χαρά θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε τώρα. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, Ε, τι, μπορώ να προσθέσω. Απλώς να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, εξ ονόματος της Πολωνικής Προεδρίας. Πρέπει να πω ότι μάθαμε πολλά, διδαχθήκαμε πολλά κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο προνόμιο. Να ακούω μάλιστα και από εσά ότι και εσείς διδαχθήκατε πολλά. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το μεταφέρω στην πολωνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ που εκτιμήσατε το έργο μας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία στο μέλλον, προ όφελο της ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά παραμένει το κρίσιμο θέμα, ιδιαίτερα σε αυτές τις ε, πολύ δυσμένες περιόδους που διαρχόμαστε αυτή τη στιγμή. Ας επενδύσουμε στην ανάπτυξη, στην ε, εξέλιξη. Και εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε καλό, καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος. Χαρούμενο νέο έτος. Ευχαριστώ πολύ. E, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ναι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, ακούγοντάς σας να λέμε, να λέτε καλά λόγια για την Πολωνική Προεδρία. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε δεν θα ε, σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές υπέρ της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Well, you very indeed for joining us. Uh, we reciprocate Σας ευχαριστούμε πολύ που προσήλθατε. Σας ευχόμαστε και εμείς καλή χρονιά και σας αξίζει αυτό το διάλειμμα. Δεν ξέρω αν είδατε ότι υπάρχει ένα νέο δελτίο τύπου για τους καταναλωτές έτσι ώστε να, να πανηγυρίσουμε αυτό το φόρουμ των καταναλωτών, να το τιμήσουμε. Σας δίνω λοιπόν αντίτυπα και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να τα λάβετε. Υπενθυμίζω όσους μας παρακολουθούν από το δίκτυο ότι μπορούν να παρακολουθήσουν, να δουν αυτό το δελτίο στη χριστουγεννιάτικη έκδοση για το τι κάναμε και τι θα κάνουμε του χρόνου. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας και μπορούμε να σας αποστείλουμε και ένα αντίτυπο. Έχουμε 1737 ε, εγγεγραμμένους στο δελτίο μας, κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δίνω το λόγο στην Μπερναντέτ Βερνιό η οποία θα αναλάβει το επόμενο, τα επόμενα θέματα, γιατί εγώ πρέπει να πάω στην ακρόαση για την περιαγωγή. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Σας αναθέτω μάλλον την Προεδρία. Eh Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Για σήμερα περνάμε τώρα στην ε, έκθεση για την επιγραμμική επίλυση των διαφορών από τους καταναλωτές και θα δούμε την ανάλυση αντικτύπου από την Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζακλίν Μίνορ από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Και παράλληλα θα, εξετάσουμε τον εξοδικαστικό κανονισμό για τις διαφορές των καταναλωτών. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην Κομισιόν, μετά στο Λουί Κρέκ και μετά στην κυρία Ρόζα Τούν, η οποία λείπει τώρα αλλά θα επανέλθει, και μετά στους Σκιώδης. Το λόγο έχει η Κομισιόν, η κυρία Ζακλίν Μινόρ. Merci, Madame la Présidente. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας παρουσιάσει σήμερα την αξιολόγηση αντικτύπου για τις δύο προτάσεις ε, που εγκρίθηκαν στις 29 Νοεμβρίου. Η πρώτη ήταν μια πρόταση οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και η δεύτερη μια πρόταση κανονισμού για την ε, επιγραμμική επίλυση διαφορών. Όπως θα γνωρίζουν περισσότεροι από εσά, ε, αυτές είναι σημαντικές δράσεις για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά, ιδίω ε, για τα ψηφιακά, για τη διαδικτυακή αγορά και ιδίω ε, για διαμεθοριακές αγορές και πωλήσει. Ο στόχος μας με αυτές τις νέες προτάσεις είναι να δώσουμε στους καταναλωτές ένα αποτελεσματικό μέσο όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν προβλήματα με αγαθά υπηρεσίες ε, με κάποιον εμπορευόμενο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο εμπορευόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν αγόρασαν τα αγαθά, είτε σε ένα κατάστημα είτε στο διαδίκτυο ε, και ανεξάρτητα από το ποια ήταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Αυτό που θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχής είναι ότι όταν ε, αναφερόμαστε στην επίλυση διαφορών, αναφερόμαστε στις εξοδικαστικές επίλυσεις διαφορών και τίποτα από αυτά που θα πω δεν έχει κάποια επίπτωση στο δικαίωμα είτε του καταναλωτή είτε του πολιτή να προσφύγει στα δικαστήρια για επίλυση διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια κοινή αξιολόγηση αντικτύπου και για τις δύο προτάσεις. Αυτά λοιπόν που σας ε, λέω ε, βασίζονται και στις δύο ε, προτάσεις, εκτός και αν διευκρινίζω ότι αναφέρομαι είτε στο ένα είτε στο άλλο. Τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης αντικτύπου ήταν τα εξής. Εξετάσαμε πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Είδαμε τι προκλήσεις, τι προβλήματα, τι ελλείψεις έχει η κατάσταση επί του παρόντος. Εξετάσαμε τις απόψεις των ενδιαφερομένων και θα θυμάστε ότι οργανώσαμε χάρη σε αυτή την επιτροπή και μια πολύ επιτυχία ακρόαση για την εναλλακτική επίλυση διαφορών πριν από 9 περίπου μήνες. Είδαμε και την αρχή της επικουρικότητας ε, με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο για τον τρόπο παρέμβασης ε, και αναλύσαμε και τις διάφορες δυνατότητες που έχουμε από πολιτική σκοπιά και επιλέξαμε μια συγκεκριμένη ως την προτιμόμενη λύση και εξετάσαμε περισσότερο εις βάθος τι επιπτώσεις έχει. Ε, η κατάσταση λοιπόν για την αναλλακτική επίλυση διαφορών. Επί του παρόντος νομίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 750 ε, διαφορετικοί φορείς εναλλακτική επίλυση διαφορών, αλλά από τη μελέτη που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσα να παρεπέμβονται και πιο πρόσφατες έρευνες που λένε ότι έχουμε πάνω από χίλια εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε εξ αρχή είναι ότι ε, διαφέρει πολύ η εναλλακτική επίλυση διαφορών από κρατο μέλος σε κράτο μέλος και είναι και πολύ διαφορετική ανάλογα με τον ε, κάθε τομέα. Και ε, την ονομάζουμε με διάφορα ονόματα. Ε, στα γαλλικά τη λέμε mediation, διαμεσολάβηση, κάτι το οποίο συγχαίει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, διότι mediation στα αγγλικά αναφέρεται σε κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο η επίλυση διαφορών. Μπορεί να είναι μια μορφή διαιτησίας, μπορεί να είναι μια μορφή ε, όπου κάποιος τρίτος προσπαθεί να συμφιλειώσει τον εμπορευόμενο και τον καταναλωτή. Μπορεί να είναι και ένα ε, ε, σύστημα επίλυσης διαφορών ή ένα σύστημα κατάθεσης αναφοράς ή παραπώνων. Ανάλογα με το κράτος μέλος λοιπόν διαφέρει ε, ακόμα και η ονομασία και θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το καθένα από αυτά ήταν μοναδικό και έχει διαφορετικούς κανόνες και μπορούν να καθοριστούν με διαφορετικό τρόπο. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη αυτά τα συστήματα επίλυσης διαφορών έχουν ε, ε, προκύψει κατόπιν όθησης από τις δημόσιες αρχές, σε κάποια άλλα κράτη-μέλη έχουν προκύψει ως πρωτοβουλία του κλάδου, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ ενός εμπορικού τομέα και μιας οργάνωσης καταναλωτών ή μιας δημόσιας αρχής που δρά ως ε, χορηγός εντός εισαγωγικών ε, σε μια τέτοια οργάνωση. Η χρηματοδότηση είναι επίσης πολύ διαφορετική ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα ε, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ε, του κάθε προγράμματος και του κάθε κράτους μέλους. Κάποιες φορές χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κλάδο, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προέρχεται αποκλειστικά από το δημόσιο κορβανά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένα αμάλγαμα των δύο και ε, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι φορείς επίλυσης διαφορών ε, χρεώνουν κάποια τέλη, κάποια αμοιβή ε, για την επίλυση της διαφοράς. Υπάρχουν επίσης κάποια προγράμματα τα οποία είναι εθνικής φύσεως και καλύπτουν όλη την επικράτεια ενός κράτους μέλους, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι περιφερειακά, ιδίως σε κράτη-μέλη που έχουν ομοσπανδιακή δομή, και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία μπορεί να είναι και τοπική φύσεω και να αφορούν μια συγκεκριμένη πόλη, ή ένα συγκεκριμένο δήμο. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι και ε, ε, υπάρχουν και συστήματα επίλυσης διαφορών και ανακλάδο αλλά και πολυτεμοιακά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές μεγάλες διαφορές αλλά υπάρχουν και κάποιες κοινέ πτυχές ε, που καλύπτονται και διαθέτουν όλα τα εθελοντικά συστήματα ε, συγγνώμη, όλα τα συστήματα. Καταρχά έχουμε την εθελοντική φύση. Όλα προκύπτουν από το κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ορισμένες φορές ε, μπορεί να είναι και ε, η προθυμία αυτή, η διάθεση να δεχτούμε αυτό το εναλλακτικό σύστημα για όποια διαφορά προκύψει. Πολλοί εμπειρευόμενοι λοιπόν δεσμεύονται να δεχτούν τη χρήση ενός συγκεκριμένου φορέα επίλυσης διαφοράς για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μεταξύ των και των πελατών τους. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ε, αντίθετα, οι εμπορευόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν αναπερίπτωση εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, την αναλλακτική επίλυση διαφορών. Επιπλέον, το αποτέλεσμα μια διαδικασία επίλυσης διαφορών είναι διαφορετικό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό, επομένως σε κάποιες περιπτώσεις αν συμφωνήσει κάποιο, να έχουμε μια εναλλακτική επίλυση διαφοράς και οι δύο φορεί ή ο εμπορευόμενο δεσμεύονται από το αποτέλεσμα. Όποια και αν είναι η απόφαση ή η σύσταση συμφωνούν να την ακολουθήσουν. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει είναι απλώ μια σύσταση. Τέλος, Κάτι το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι ελάχιστα από τα υφιστάμενα προγράμματα ασχολούνται αποκλειστικώ και μόνο με τις διαδικτυακές αγορές. Υπάρχουν κάποια ε, λίγα ε, κάποιες λίγες περιπτώσεις συγγνώμη, που αφορούν ε, διαδικτυακές αγορές. Κάποιες έχουν κάποιο εγκεκριμένο τομέα που ασχολείται με το διαδίκτυο, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για τις διαδικτυακές αγορές και είναι ελάχιστοι αυτοί που διαχειρίζονται την όλη διαδικασία διαδικτυακά. Ακόμα και αν αγοράσετε τα αγαθά σας δηλαδή από το διαδίκτυο, μπορεί να πρέπει να πάτε σε ε, κάποιο ε, φορέα αναλλακτικής επίλυσης διαφορών τύπου bricks and water. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία είναι κοινά, το ότι είναι επιθελούσιας βάσεως, όλα αυτά γίνονται εξοδικαστικά και υπάρχει παρέμβαση ε, κάποιου τρίτου φορέα. Ακόμα και αν ο τρίτος ε, φορέας ε, μπορεί να κάνει απλώς και μόνον την επαφή μεταξύ εμπορευόμενου και πελάτη προκειμένου να συνεννοηθούν και να καταλάβουν καλύτερα ποια είναι η διαφορά τους. Όλα αυτά σημαίνουν βέβαια ότι η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι πιο γρήγορη, είναι λιγότερο δαπανορή και είναι και φυσικά απλούστερη για την επίλυση διαφορών από ότι θα ήταν μια δικαστική διαδικασία. Και αν μιλήσετε και με τους καταναλωτές αλλά και με τους εμπορευομένους, αυτοί που έχουν πείρα εναλλακτική επίλυση διαφορών τη βλέπουν ως κάτι πολύ θετικό. Όταν μιλούμε λοιπόν με τους καταναλωτές ε, για την ε, προετοιμασία της ε, αξιολόγησης αντικτύπου, αυτοί που τη χρησιμοποίησαν τη θυμούνται κάτι κάτι απλό, ε, καθόλου περίπλοκο, μπόρεσαν να λάβουν ε, κατάλληλες συμβουλές και γνώμες από τον αντίστοιχο φορέα και ε, συνήθως έλυσαν το πρόβλημά τους. Ε, και στις επιχειρήσεις το 73% δηλαδή τα 3 τέταρτα αυτών που χρησιμοποίησαν την ελλακτική επίλυση των διαφορών ήταν ικανοποιημένοι και ένα 82% 8 στους 10 δηλαδή δηλώνουν ότι θα την ξαναχρησιμοποιούσαν στο μέλλον. Και μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, το 70% λένε ότι θα προτιμούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μορφή επίλυσης διαφορών από το να προσφύγουν στο δικαστήριο. Οι ελλείψεις τώρα. γιατί θεωρήσαμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά ως υπόβαθρο, υπάρχει λόγος να το εξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαπιστώσαμε τέσσερα κύρια μειονεκτήματα. Το πρώτο ήταν κάποια κενά στην κάλυψη της εναλλακτική επίλυσης διαφορών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα, περίπου μεταξύ 750 και 1000 προγράμματα επίλυσης διαφορών, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση διαφορών όταν υπάρχει διαφορά με έναν, ε, με έναν εμπορευόμενο. Υπάρχουν κενά ε, και αναχώρα και ανατομέα. Και αν δείτε λίγο την αξιολόγηση αντικτύπου υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που είναι τα προ... πια προφανή κενά. Ε, θα τα δείτε αυτά και μέσα στο κείμενο και στα παραρτήματα. Στην πράξη λοιπόν οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν επιλύουν τις διαφορές τους με τους εμπορευομένους. Ε, απευθύνονται στον εμπειροβόμενο. Οι περισσότεροι καταναλωτέ, όταν έχουν ένα πρόβλημα με αγαθά ή υπηρεσίε που αγόρασαν, είτε πηγαίνουν στο κατάστημα, είτε στην ιστοσελίδα από όπου αγόρασαν ε, κάτι, ε, και όταν δεν έχει αυτό αποτέλεσμα, οι περισσότεροι παρετούνται. Απλώς δέχονται ότι έχασαν ε, σε αυτή την περίπτωση και ο υπολογισμός ο οποίος δίνεται αναλυτικά στην αξιολόγηση αντικτύπου υποδηλώνει ότι το 0,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αντιστοιχεί στις απώλειες που έχουμε ε, λόγω ε, προβλημάτων στην επίλυση διαφορών. Πολλοί καταναλωτές λοιπόν όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις αγορές τους δεν τις επιλύουν. Και αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα στους καταναλωτές, γι' αυτό είναι σαφές, αλλά και για τις καλές επιχειρήσεις. Διότι ε, αυτά είναι κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ταπανίσει καταναλωτές σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες από ε, πιο υπεύθυνους εμπορευμένους. Όσον αφορά τώρα τα κενά, ξέρουμε ότι ιδίω σε δια... μεθοριακό επίπεδο υπάρχουν προβλήματα. Πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών, γιατί δεν μπορούν να βρουν κάποιον στον οποίο μπορούν να αποτανθούν στη χώρα του εμπορευομένου οι καταναλωτές. Δεύτερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν είναι τόσο γνωστή η εναλλακτική επίλυση διαφορών περίπου το 30% των Ευρωπαίων καταναλωτών δεν έχουν ακούσει ποτέ την ύπαρξη ε, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δεν ήξεραν ε, τίποτα για αυτόν τον τρόπο ε, επίλυσης της διαφορές τους και 40% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, οι μισές περίπου ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν ε, φορείς ή προγράμματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με τα οποία θα μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματά τους. Το τρίτο πρόβλημα που εντοπίσαμε ήταν η ποιότητα των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1998 και το 2001 ενέκρινε κάποιες συστάσεις που καθόριζαν κάποιες βασικές αρχές οι οποίες κατά την άποψή μας θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις ε, εναλλακτικές επιλύσεις εφορών. Ε, στοιχεία που αναφέρονται στην ε, διαφάνεια, στην αντικειμενικότητα και ούτω καθεξής. Αυτές βεβαίως είναι συστάσεις, δεν είναι δεσμευτικές και ε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας περίπου το 60%, κάτι λιγότερο από το 60% των ε, ε, υφιστάμενων ADR ε, τα εφαρμόζουν, που σημαίνει ότι έχουμε ένα 40% που δεν συμμορφούνται προς αυτές τις αρχές και φυσικά δεν έχουμε κανένα τρόπο να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συμμόρφωση προς αυτές τις αρχές. Κάτι επιπλέον το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι η χρήση μιας σύστασης σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνεκτική παρακολούθηση αυτών των αρχών. Δεν υπήρχε ανάγκη οι δημόσιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλο φορέας να ελέγξει ότι υπάρχει συμμόρφωση προς αυτές τις συστάσεις. Και ένα τέταρτο πρόβλημα τέλος είναι η συγκεκριμένη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά τα, ε, τις διαδικτυακές, διαμεθοριακές ε, εμπορικές συναλλαγές. Θα γνωρίζετε όλοι τα στοιχεία, διότι επαναλαμβάνονται ε, μονότανα συνεχώς ε, σε οποιαδήποτε συζήτηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 40% των Ευρωπαίων κατά μέσο όρο έχουν κάνει τουλάχιστον μία αγορά στο διαδίκτυο. Ε, τη χώρα τους, αλλά μόνο περίπου το 9% έχουν αγοράσει αγαθά υπηρεσίες από, μια ε, ιστοσελίδα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Και αυτά τα στοιχεία είναι ε, πολύ συγκεκριμένα. Ενώ η εσωτερική διαδικτή αγορά αυξάνεται πολύ γρήγορα, η διαμεθοριακή διαδικτυακή αγορά αναπτύσσεται πολύ αργά. Και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ε, κάποιοι διστάζουν να αγοράσουν ε, αγαθά σε άλλη χώρα μέλα Σίγουρα η γλώσσα ε, δημιουργεί προβλήματα, η γνώση μιας μάρκας, η φήμη ε, ενός εμπορευομένου, αλλά σχεδόν ε, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές πιστεύουν ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να επιλύσουν ένα πρόβλημα εάν προκύψει με κάποιο διαδικτυακό κατάστημα σε άλλο κράτος μέλος. Και αυτό πιστεύουν ότι θα τους δημιουργήσει και πρόβλημα για τις επισκευές ή τις αλλαγές αν το έχουν αγοράσει από κάπου εκτός ε, ε, της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το δείτε αυτό και από πλευράς εμπορευομένου είναι ακόμα πιο προφανές. Το 60% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λένε ότι είναι υψηλότερο το κόστος επίλυσης διαφορών με καταναλωτές που βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, γι' αυτό και δεν πουλούν, πουλούν σε άλλες αγορές, σε άλλα Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε τι ελλείψεις υπάρχουν. Όπως ε, ξέρετε εξετάσαμε και τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων. Έγινε μια πολύ επιτυχημένη ακρόαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε πάνω από 200 διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων που απάντησαν στην ε, διαδικασία διαβούλευσής μας. Σχεδόν όλοι συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω τα θέματα εναλλακτική επίλυση διαφορών και να υπάρχει και υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι απόψεις μας ε, τότε παρουσιάστηκαν σε μια σύνοψη στο διαδίκτυο και συνοψίζονται φυσικά και ε, στην αξιολόγηση αντιπτύπου. Υπήρχε και μια αξιολόγηση της αρχής της επικουρικότητας. Βέβαια δεν χρειάζεται να το υπενθυμίσω εδώ ε, στην Επιτροπή σας ότι στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και θα πρέπει να διασφαλίζει τα συμφέροντά τους ώστε να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτά είναι από τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όψη, κατά την άποψη τη της Επιτροπής η απουσία ενός αποτελεσματικού εναλλακτικού συστήματος επίλυση διαφορών δημιουργεί προβλήματα για την επίλυση διαφορών στους καταναλωτές στα διάφορα κράτη-μέλη, ιδίως ε, σε επίπεδο διαμεθοριακού εμπορίου και ε, φυσικά αυτό αποτελεί πρόσκομα για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια αποτελεσματικά ε, λειτουργούσα ε, δομή αποτελεσματικό και καλά λειτουργών σύστημα επιλυση διαφορών θα πρέπει να δημιουργηθεί σε ένα αποτελεσματικό και καλά λειτουργών σύστημα επίλυσης διαφορών σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να έχουμε διασυνοριακό σύστημα επίλυσης διαφορών εάν δεν έχουμε ένα δίκτυο ε, εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών σε εθνικό επίπεδο. Και το συμπέρασμά μα ήταν ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να προάγουμε το ίδιο επίπεδο προστασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Να δούμε τώρα τι επιλογές έχουμε από πλευράς πολιτικής πολύ γρήγορα. Η πρώτη επιλογή ήταν να μην γίνει τίποτα για το εναλλακτικό σύστημα επίλυση διαφορών, να αφήσουμε τα πράγματα ως όχουν και να βασιστούμε απλώς και μόνο στη φυσική εξέλιξη του συστήματος ε, μαζί με τα κίνητρα ε, βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουμε ήδη ενισχύει. Η δεύτερη δυνατότητα ήταν να συνεχίσουμε με τη μη δεσμευτική προσέγγιση, δηλαδή να επικαιροποιήσουμε τις συστάσεις και ε, να τη συνοδεύσουμε και με καλύτερη ενημέρωση προς τους καταναλωτές ε, για το εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών. Η τρίτη λύση ήταν ένα ε, νομικό δεσμευτικό μέσο, ώστε οποιοδήποτε να μπορεί να παραπέμπει τα προβλήματά του στο ε, σύστημα επίλυσης διαφορών και να είναι και καλά ενημερωμένος ε, για την ύπαρξη αυτών των συστημάτων. Και η τέταρτη λύση ήταν να υπάρχει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο και πάλι, όπως και στην τρίτη επιλογή, αλλά σε αυτή την περίπτωση να δημιουργήσουμε μέσω αυτού του νομικού μέσου ένα κοινό ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Αυτές ήταν λοιπόν οι τέσσερις εναλλακτικέ λύσεις για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Μετά εξετήσαμε τα διαδικτυακά θέματα επίλυση διαφορών. Οι δύο πρώτες εναλλακτικέ λύσεις ήταν και πάλι οι ίδιες, να μην γίνει τίποτα ή να δράσουμε μόνο μέσω ενός μη δεσμευτικού μέσου ε, ενιδησίστασης. Η τρίτη επιλογή που εξετάσαμε ήταν μια δεσμευτική λύση από νομική σκοπιάς, η μορφή της οποίας θα ήταν να δρασουμε μονο μεσω ενος μη δεσμευτικου μεσου συσταση η τριτη επιλογη που εξετασαμε ηταν μια δεσμευτικη λυση απο νομικη σκοπιας η μορφη της οποια θα ηταν να εχουμε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών, να έχουμε δηλαδή ένα κόμβο ε, και η τελευταία, η πιο ακραία που εξετάσαμε, ήταν να δημιουργήσουμε ένα κανονισμό ο οποίος θα καθορίζει έναν ενιαίο φορέα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών. Θα υπάρχει δηλαδή ένας φορέας ε, διαδικτυακής επίλυσης ε, με προσωπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ασχολείται με τα θέματα αυτά πανευρωπαϊκά. Αυτό που αποφασίσαμε ε, τώρα ως καλύτερη λύση ήταν ότι εάν δεν υπήρχε καμία ευρωπαϊκή δράση, τα πράγματα θα εξελιχθούν. Όλοι πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν ούτως ή άλλως, αλλά ε, πολύ αργά και μπορεί και να μην είναι και τόσο ικανοποιητικά όσο ε, θα ήταν αν είχαμε και την ε, ε, όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάσαμε και τα μη δεσμευτικά μέσα, αλλά νομίζουμε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι και τόσο σημαντικές και Απορρίψαμε την τέταρτη επιλογή και στις δύο περιπτώσεις, ενός ενιαίου μοντέλου εναλλακτική επίλυση ε, διαφορών και ενός ενιαίου φορέα διαδικτυακών ε, ε, διαφορών, διότι θεωρήσαμε ότι δεν θα τηρείται επικουρικότητα και θα υπάρχει και πολύ μεγάλο επιπλέον άχθος. Ε, επιλέξαμε λοιπόν την τρίτη λύση, ένα δεσμευτικό μέσο για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, ώστε να καλύψουμε τις ελλείψεις για την κάλυψη και την ποιότητα των πληροφοριών και ένα κανονισμό ο οποίος θα συστήνει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών που θα βασίζεται στους εθνικούς φορείς επίλυσης διαφορών. Καθυστερώ βέβαια, αλλά προσπαθώ να τελειώσω την παρουσίαση ε, της αξιολόγησης αντικτύπου και μετά θα σταματήσω. Γιατί θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αυτή η τρίτη λύση η καλύτερη λύση. Γιατί ο στόχος μας ήταν πάντα να έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές όπου και αν βρίσκονται σε ένα ποιοτικό φορέα επίλυσης διαφορών. Και θεωρούμε ότι ο συνδυασμός οδηγίας και κανονισμού θα το προσφέρει αυτό στους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ακόμα και 20 δισεκατομμύρια ετησίω. και επίσης θεωρούμε ότι θα είναι και μεγάλο το όφελος για τις επιχειρήσεις με τη χρήση αυτού του εναλλακτικού συστήματος επίλυσης διαφορών. Και αυτό προέκυψε σαφώς και στο φόρουμ της ενιαίας αγοράς στην Κρακοβία, διότι βελτιώνει τη φήμη των επιχειρήσεων, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντλήσουν διδάγματα από αυτά τα οποία βλέπουν από τα προβλήματα και τις διαφορές οι οποίε είναι εξελίξει στα συστήματα επίλυση διαφορών και πιέζοντά του να είναι πιο υπεύθυνοι ή ενθαρρύνοντά του, αν θέλετε, να είναι πιο υπεύθυνοι για τα προβλήματα των καταναλωτών, γίνονται πιο αποτελεσματικοί και πιο ανταγωνιστικοί. υπολογίσαμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξοικονοποιήσουν ε, αρκετά μεγάλο ποσά. Είναι δύσκολο να κάνουμε ακριβή εκτίμηση, αλλά θεωρούμε ότι το ελάχιστο θα είναι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το αναφέρουμε στην αξιολόγηση αντικτύπου και μπορεί να φτάνουμε μέχρι και στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό είναι το κόστος που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε ε, Εάν ε, δεν προσφύγει κάποιο στο δικαστήριο, θα είναι και εξοικονόμηση χρημάτων όταν ε, διορθώνεται η κατάσταση και δημιουργείται μια καλύτερη φήμη για την επιχείρηση. About... Δύο λόγια σχετικά με το κόστος, διότι κάποιες χώρες μέλη βεβαίως λαμβάνουν και αυτό υπόψη και το βάρος, το οικονομικό για τη θέσπιση φορέων ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Βεβαίω, είναι πολύ δύσκολο να το μετρήσει κανεί, εξαρτάται από το εύρος και το πεδίο το ε, εδαφικό και ως προς το περιεχόμενο. 100.000 ε, πούμε ευρώ χρειάζονται για την θέσπιση ας πούμε αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο ας πούμε κόστισε πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο, διότι υπάρχει ένας διαμεσολαβητής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, ένας ombudsman. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται αυτοί οι φορείς, ADR, ε, θα αποφασιστούν από τις χώρες μέλη. Όταν ρωτάμε τις επιχειρήσεις, το 60% απάντησαν ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του φορέα. Πέρα λοιπόν από το κόστος, το άλλο κόστος είναι η ενημέρωση πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στην οδηγία. Το κόστος αυτό εκτιμάται 200-250 ευρώ ανά επιχείρηση, δηλαδή το να βάλει κανείς τις πληροφορίες, τα τιμολόγια, στις αποδείξεις και στο ε, ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα. Ε, βέβαια για, για μια εμπορική επιχείρηση δεν νομίζουμε ότι είναι πολύ ψηλό αυτό το κόστος. Τώρα, βεβαίως η πλατφόρμα, η δημιουργία της πλατφόρμας είναι δουλειά της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και 300.000 θα είναι η ετήσια συντήρηση. Και βεβαίως θα υπάρχει και το κόστος των εμπειρογνωμόνων και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Ίσως πρέπει να σταματήσω εδώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες και τις ερμηνείες. Ασφαλώς θα χρειαστεί χρόνος, διότι είναι πράγματι θέματα που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Θα δώσω το λόγο στους ε, βουλευτές και στους συγητές. Θα δώσω το λόγο στον Λουίς Κρέσιο και μετά στην κυρία Τούν και στη συνέχεια δεν ξέρω αν η η Ιβάνοβα είναι εδώ, όχι, Μήτρο δεν είναι εδώ, αλλά και πάλι ο Λουίς μπορεί να τους εκπροσωπήσει και μετά θα δούμε. Καταρχήν δίνω το λόγο στον Λουίς. Ο Λουίς το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ την κυρία Μάινερ για την ε, ε, καθαρή και ολοκληρωμένη πρόταση της Κομισιόν. Οι προτάσεις αυτές ε, συνιστούν μια σταθερή και υγιή βάση για όλους τους Ευρωπαίους ε, καταναλωτές ώστε να υπάρξει μια ένα σύστημα εναλλακτικής επίλυσης ε, διαφορών. Ε, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα και ξέρουμε ότι αυτή η Επιτροπή πολύ συχνά μιλάει για τα κενά της εσωτερικής αγοράς σε συνδυασμό με την παρούσα κρίση που ε, ουσιαστικά εμποδίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τα κενά αυτά επισημάνθηκαν και από τη σχετική μελέτη ε, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι ε, δεν εφαρμόζονται ε, τα όσα συμφωνούνται και υπάρχει έλλειψη ενός συστήματος συντονισμού. Η μη ύπαρξη εναλλακτικών φορέων, ε, μάλλον φορέων εναλλακτικής επίλυσης ε, διαφορών, ουσιαστικά υπονομεύει την εσωτερική αγορά και είναι καιρός πλέον τα ADR, οι φορείς αυτοί, να γίνουν ένα στις κανονικές φορές που θα εξυπηρετεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι σαφής και συνεκτική και δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες, ιδιαίτερα στα άρθρα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις και τα ADRs να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα ε, προγράμματα και τις διαδικασίες. Τίποτα δεν θα χρησιμοποιηθεί αν δεν είναι ενημερωμένοι οι καταναλωτές. Δηλαδή, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών, αλλά δεν διαθέτει επαρκή ενημέρωση του κοινού. Υπάρχουν όλα τα συστατικά στοιχεία, αλλά κάποια σημεία χρειάζονται διευκρίνηση. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να εξεταστεί. Οι Κομισιόν και οι χώρες μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ανεξάρτητα από το πώς θα χρηματοδοτηθεί το σύστημα θα πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα ανοιχτά και με διαφάνεια. Επαρκείς εξασφαλίσεις θα πρέπει να υπάρχουν ώστε να μην υπάρξουν απαιτήσει από ε, την υπονόμευση των συστημάτων εναλλακτική επίλυσης ε, διαφορών. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση. Πρέπει να δούμε ποιο θα είναι αυτό το διάστημα. Επίσης θα ήθελα η Κομισιόν να προχωρήσει πέραν ε, του καθορισμού των αρμοδιοτήτων σε κάθε χώρα μέλος. Θα πρέπει να ηγηθεί και στο συντονισμό την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και τη διάδοση των ε, απαραίτητων πληροφοριών. Ελπίδα μου είναι ότι θα έχουμε νομοθεσία στα προσεχή χρόνια που μαζί με τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα ολοκληρώσουν την προσπάθεια. Τελειώντας κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να πω ότι η εμπιστοσύνη του κοινού είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και πιστεύω ότι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης. Το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές ότι πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρωτοβουλία όπου θα πρέπει να ε, θέσουμε στον ε, νέο μηχανισμό της εσωτερικής αγοράς, στη διάθεση του μηχανισμού της εσωτερικής αγοράς, τα ADRs, δηλαδή τα συστήματα εναλλακτικής επίρρησης διαφορών και να πω τελειώνοντας ότι αυτό είναι πολύ καλό και για τους πολίτες και καταναλωτές, αλλά και επειδή συμβάλλει στο να γίνει η ενιαία αγορά πραγματικά ενιαία. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ροζατούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Συγχαρητήρια στην κυρία Μάινορ και όλη της την ομάδα. Ε, δείχνει να είναι ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός, προς την πρόοδο. Και αναμένω τη συνεργασία των προσεχή μήνα και για τα ADRs και για τα ODRs, δηλαδή και για τις εναλλακτικές ε, τους φορείς εναλλακτικής επίρρησης διαφορών και για τη διαδικτυακή επίρρηση διαφορών, ODR. Συμφωνώ επίσης ότι η πληροφόρηση σχετικά με τα εργαλεία αυτά πρέπει να είναι αποτελεσματική. Πολύ καλύτερη από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα, διότι οι πάντες παραπονιούνται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για γοργότερη οικονομική ανάπτυξη που χάνεται. Πιστεύω ακράδατα ότι αν, αν δημιουργήσουμε μια τέτοια πλατφόρμα ODR, δηλαδή για διαδικτυακή επίλυση διαφορών. Ε, πιστεύω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Ε, βέβαια ασχολούμαστε με ένα ε, τέτοιο ε, θέμα την παραμονή των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ίσως όμως είναι και πολύ χρήσιμο γιατί θα το έχουμε στο μυαλό μας καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών και θα δώσει νέα όθηση στις εργασίες μας το προσεχές έτος. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ανακοινώνεται η διαβούλευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάνω από 200 διαφορετικές ομάδες απάντησαν. Πόσα άτομα πόσα άτομα απάντησαν και αν αυτές οι διαβουλεύσεις, η ανταλλαγή απόψεων έγινε και στις 23 γλώσσες ή αν έγινε σε δύο ή τρεις όπως γίνεται συνήθως από πλευράς Κομισιόν. Διότι η διαβούλευση είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε οπωσδήποτε αν θέλουμε τα νέα κομισιων διοτι η διαβουλευση εργαλεία πραγματικά να αποδώσουν, αν θέλουμε να διευκολύνουμε πραγματικά τη ζωή των πολιτών και δεν προσθέτουμε απλώς καινούργια ονόματα, καινούργια, καινούργια βάρη πάνω επί της κεφαλής των πολιτών. Δεν θέλω να επισέλθω σε τεχνικούς όρους και θέματα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι η σε βάθος συζήτηση θα διεξαχθεί όταν σημειωθεί πρόοδος στο θέμα των ε, ADR, γιατί εκεί θα βασιστεί και το ODR. Άρα λοιπόν σταματώ εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιβάνοβα δεν είναι εδώ, άρα λοιπόν δίνω το λόγο στον κύριο Σάπο, ο οποίος το έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Μάιερ είναι ο σκιώδης νομίζω. Και ο κύριος Μάιερ είναι εδώ. Άρα λοιπόν μπορεί να λάβει το λόγο αυτός. Es tut mir leid, ich habe noch äh, wichtige Besuchergruppen hier. Όπως ξέρετε, είχα ένα μεγάλο ρυθμό επισκεπτών που συνόδευσα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε μία πρόταση οδηγίας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς ορίζεται γενικότερα η πρωτοβουλία. Εάν λάβουμε υπόψη τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία απλή λύση, να έχουμε να κάνουμε με ένα εθελούσιο σύστημα και αυτό το ανέφερε και η Πολωνική Προεδρία. Θα πρέπει να είναι ορθολογικό και οικονομικό. Θα πρέπει να προβεί σε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα τεχνικά ζητήματα ομοιόμορφα στα κράτη-μέλη. Μιλάμε για 750 με 1000 εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι συλλογικές προσφυγές δεν έχουν να κάνουν κάτι με την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Πρόκειται για μία εξοδικαστική διαδικασία. Πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό με τις ε, μαζικές προσφυγές. Σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε τα εξής. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα. Πώς μπορούμε να υποπτεύσουμε όπως θέλει η Κομισιόν. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο. Τη στιγμή που υπάρχει ε, μία παραβίαση της οδηγίας. Δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει απολυθεί. Επίσης, ε, μιλάμε για την υποστήριξη των κρατών μελών, έτσι ώστε να επιληθούν αυτές οι διαφορές. Το θέμα αυτό οδηγεί σε συγχύσεις και πρόκειται για ένα μηχανισμό γραφειοκρατικό και πολυδάπανο. Τώρα, ως προς την χρηματοδότηση θα πρέπει να διασαφινιστεί το ζήτημα στα 27 κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να το ορίσουμε σε σχέση με την εναλλακτική επίλυση διαφορών, διότι εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Θα πρέπει να υπηρετήσουμε τους καταναλωτές. Θα ήθελα να πω στην Κομισιόν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ξέρουν τις δυνατότητες που προϋπάρχουν, δηλαδή θα πρέπει να γίνει μία εκστρατεία πληροφόρησης θα πρέπει να γίνει μία εκστρατεία πληροφόρησης η οποία να είναι συστηματική και από πλευράς Επιτροπής και από πλευράς κρατών μελών. Θα πρέπει να συνεργαστούν εκ του Γιατί και οι καλύτερες διαδικασίες δεν θα υπηρετήσουν τίποτα αν δεν τις γνωρίζουν οι καταναλωτές οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν το μηχανισμό της εναλλακτική επίλυσης διαφορών και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα. Εάν μία επιχείρηση θέλει να συμμετάσχει, θα πρέπει να ξέρει πώς, θα έχει, πώς μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα. Γι' αυτό χρειάζεται μία εκστρατεία πληροφόρησης. Υπάρχουν και άλλα θετικά ζητήματα δηλαδή ο μηχανισμός εποπτείας όταν υπάρχουν ε, περιορισμένες αξιώσεις και όταν κανείς απευθύνεται σε ένα δικαστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση, δηλαδή κάθε δικαστήριο θα πρέπει να έχει κάποιον ο οποίος να γνωρίζει τον νόμο το γράμμα του νόμου υπέρ των καταναλωτών, διότι αυτό δεν το βλέπουμε ούτε στη Γερμανία. Όταν εγώ ρώτησα του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μου είπαν ναι, στέλνουμε μία εγκύκλιο στα δικαστήρια και θα πρέπει τα δικαστήρια να δράσουν αναλόγως. Δεν γίνεται όμως έμπρακτα αυτό, ούτε στη Γερμανία. Γι' αυτό σας προτρέπω να προωθήσετε μία εκστρατεία πληροφόρησης και να εξετάσετε πώς μπορείτε να θέσετε σε εφαρμογή αυτή την πλαισίωση. Πέρα από τις εκστρατείες πληροφοριών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα προαιρετικό σύστημα, ανεξάρτητα με το πώς ονομάζεται. Δηλαδή δεν ε, πρέπει να πρόκειται για μία εξοδικαστική οδό η οποία αποκλείει την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικό. Θα πρέπει κανείς να μπορεί να προσφύγει με αγωγές και στα εθνικά δικαστήρια. Απλώς διασαφηνίζει κάπως τα πράγματα και είμαι πεπισμένος ότι οι εισηγητές και ιδιαίτερα οι σκιώδεις θα μπορέσουν να συνεργαστούν επί του θέματος. Alors, je vais donner la euh, Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις τώρα. Ο ε, κύριος Ρέπο δεν είναι εδώ. Από πλευρά σοσιαλιστών νομίζω ε, ότι ο Λουίς θα πάρει το λόγο. Ναι, εξ του κυρίου ε, Ρέπο. Ναι, και εξ ονόματός σας. Ο κύριος Ρέπο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γι' αυτό μιλώ εξ ονόματός του. Σας διαβάζω τη σημείωσή του. Καλωσορίσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπε ότι θα, μετά το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει ε, διευρυνθεί και η ηλεκτρονική αγορά διασυνοριακά, όμως είναι δύσκολο να υπάρχουν διασυνοριακές συναλλαγές γιατί φοβούνται οι καταναλωτές ότι δεν μπορούν να επιληθούν διαφορές διασυνοριακώς. Γι' αυτό ο κύριος Ρέπο θεωρεί ότι όλα τα μέτρα που προωθούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά είναι ύψης της σημασίας. Γι' αυτό προτείνει μία πλατφόρμα, μία επιγραμμική πλατφόρμα για όλους τους αγοραστές, έτσι ώστε να διαδίδονται αυτές οι προπτικές. Τα σημεία εισόδου θα πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήση, προσβάσιμα και σε όλες τις γλώσσες, καθώς και χωρίς δαπάνη θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες στα εμπλεκόμενα μέρη έτσι ώστε να υπάρχει ίση πρόσβαση στους καταναλωτές και στους εμπόρες. Υπάρχουν Υπάρχουν όμως και προκλήσεις από πλευράς διαδικτυακής επίλυσης διαφορών. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες που να διέπουν τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών, να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλες τις ομάδες, ακόμα και τις πιο ευάλωτες υψηλή ποιότητα ασφάλειας στο διαδίκτυο καθώς και δυνατότητα χρήσης του συστήματος. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα βοήθεια στη μητρική γλώσσα του καταναλωτή να μην επιβαρύνονται αυτές οι υπηρεσίες και να υπάρχει ουδετερότητα της διαδικασίας διαδικτυακής επίλυσης διαφορών. Ο κύριος Ρέπο ελπίζει να συνεργαστεί με τον εισηγητή και άλλους επί του θέματος αυτού. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν. Να μιλήσει καταρχήν ο κύριος Σφάμπ γιατί πρέπει να φύγει. Είπα ότι πρέπει να φύγετε κύριε Σφάμπ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο κύριος Μάγερ ήδη είπε αρκετά, έθιξε αρκετά ζητήματα. Είπε ότι θα πρέπει να είναι ένα εθελούσιο σύστημα, ένα μη δεσμευτικό σύστημα. Και ως προς την πληροφόρηση είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ συλλογικών αγωγών και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής ε, τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του. Το εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών δεν είναι γνωστό ούτε στον καταναλωτή ούτε στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε οικονομικές λύσεις χωρίς να πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Το Bundestag ενέκρινε αυτές τις ε, μέρες ένα σύστημα διαιτησίας μέσω ειρηνοδικών. Και αυτό μπορεί να γίνεται επιγραμμικά ή όχι. Θα πρέπει όμως να υπάρχει εμπιστοσύνη. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε κανόνες για την προώθηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή, γιατί πρέπει όχι μόνο να γνωρίζει το σύστημα, αλλά να του έχει και εμπιστοσύνη. Μιλάμε για την προσφυγή σε ένα δικαστήριο για να μπορέσει να προωθήσει τα δικαιώματά του. Εάν ήταν δεσμευτικό αυτό το σύστημα, τότε θα μπορούσε άμεσα να προσφύγει σε ένα δικαστήριο. Πρόκειται για μία προγενέστερη φάση πριν κανείς προσφύγει στη δικαιοσύνη δηλαδή. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσουν και οι δύο διαδικασίες πώς να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή έτσι ώστε να ελαφρύνουμε και τα δικαστήρια και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τα δικαιώματά του σε μία διαδικασία επίλυσης. Ως προς το επιγραμμικό σύστημα μπορούμε κάτι να κάνουμε υπέρ της ενιαίας αγοράς. Γιατί εάν μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το σύστημα επίλυσης των διαφορών επιγραμμικά, τότε θα αυξηθεί και η εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές συναλλαγές, κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι τώρα. Έτσι θα φτάσουμε σε μια πραγματική ενιαία αγορά. Εάν λοιπόν Μπορεί κανείς online να επιλύσει διαφορές με μία επιχείρηση, που να προβάλλει και τα δικαιώματά του και να εμπιστευτεί το σύστημα. Μπορεί δηλαδή να προβάλλει τα αιτήματά του έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αμελητοί. Νομίζω ότι και οι δύο διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές για την εκ νέου εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ενιαία αγορά και θα ήθελα ο εισηγητής και οι σκιώδεις να εξετάζουν πώς μπορεί να επιταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών για να τους προστατεύσουμε. Πώς λοιπόν οι καταναλωτές πριν προσφύγουν στη δικαιοσύνη πριν προβούν σε μια συλλογική αγωγή ή προσφυγή, να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τα δικαιώματά τους μέσω αυτής της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που προελέχθησαν. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι Τούν και Μάιερ. Νομίζω ότι η Επιτροπή ευτυχώς προέβαλε μία ε, οδηγία, μία πρόταση οδηγίας για να ισχύσει μακροχρόνια και με μία πολύ σταθερή βάση. Τι, τις περισσότερες λεπτομέρειες τις γνωρίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι εξαιτίας αυτών των προπαρασκευαστικών διεργασιών μπορούμε να φτάσουμε σε διαβουλεύσεις. Δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει το Μάρτιο, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε έναν οδικό χάρτη για να δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να γίνει μια ακρόαση και ενδεχομένως πότε. Και πότε θα έχουμε την πρόταση έκθεσης. Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ο επιχειρηματικός κόσμος τάσεται υπέρ της πρότασης αυτής. Κατά πόσο θεωρεί ότι αυτή η πρόταση παρουσιάζει ενδιαφέρον ή κατά πόσο θα πρέπει να προβάλλουμε τροπολογίες. Όπως είπε και ο Hans Peter Mayer, το σύστημα θα λειτουργήσει εάν υπάρχουν οι σωστές, η σωστή πληροφόρηση για την διαδικασία. Γιατί πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί σκλήρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πραγματικά αυτό το πλαίσιο. Αυτή η ανταλλαγή είναι πολύ επικοδομητική και θα το συνεχίσουμε ως σκιώδης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δράσουμε με σπουδή. Η κυρία Γκέπχαρτ δεν είναι παρούσα. Θα πρέπει όμως να ξαναδούμε αυτή την πλαισίωση και να ε, περάσει το θέμα πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Να περάσει στην Ολομέλεια και να εγκριθεί από αυτήν. Εγώ παρουσίασα ε, τα δεδομένα αυτής της συζήτησης. Δεν μπορούμε να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει, υπάρχουν, περίπου 20, υπάρχουν περίπου 20 σημεία που θα μας απασχολήσουν τον Ιανουάριο. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν οδικό χάρτη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν που μας παρουσίασε το θέμα τόσο διεξοδικά. Ήταν διεξοδική η παρουσίαση και θεωρώ ότι η πρόταση είναι, η αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανέξοδη. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο που βρίσκεται αυτή η πρόταση έτσι ώστε να ευεργητεί πραγματικά και τους καταναλωτές και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα τεθεί το θέμα στην Κομισιόν. Ευχαριστούμε κυρία Σφαμπ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο μεταξύ των παρεστομένων βουλευτών. Όχι. Επομένω. θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Πολωνική Προεδρία, στον κύριο Πάβελ Σαγκάη. Είπαμε όλοι και πολύ ειλικρινά ότι η Πολωνική Προεδρία έλαβα αποφάσεις που ήταν πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες. 13 ε, και 14 Δεκεμβρίου είχατε αυτή τη τόσο σημαντική έκθεση για το θέμα αυτό και σας δίνω απευθεία το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο εδώ. Γι' αυτό και θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους παρισταμένους σε αυτή την αίθουσα, ευρωβουλευτές αλλά και τους υπολείπους. Συμφωνώ απολύτως με την πρόεδρο, η οποία είπε ότι η Πολωνική Προεδρία για το θέμα αυτό, για τα προγράμματα του ΡΑΛ προσπάθησε να προχωρήσει τις εργασίες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την Επιτροπή ΙΜΚΟ, η οποία οργάνωσε με τόσο ταχύ τρόπο την πρώτη ακρόαση που σχετίζεται και με τα δύο αυτά νομοθετικά κείμενα. Διότι θέλουμε και οι δύο να εγκριθούν τα θέματα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Η συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται ότι ξεκινά ε, καλά. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Στο Συμβούλιο αφιερώσαμε τρεις μέρες εργασίας ε, για τα θέματα αυτά. 29 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και όπως είπε και η Πρόεδρος στις 13 και 14 Δεκεμβρίου ήδη ξεκίνησε μία πιο εις βάθος συζήτηση και για τα δύο αυτά ζητήματα. Και επίσης ε, ξεκινά και η συζήτηση με μία παρουσίαση της αξιολόγησης αντικτύπου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι όλες αυτές τις ε, ημέρες ε, ευθύς εξ αρχής απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες ορισμένες φορές ήταν και δύσκολες ερωτήσεις από πλευράς κρατών μελών και νομίζω ότι αυτές οι απαντήσεις μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε ποιος είναι ο στόχος ε, των νομοθετικών κειμένων. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι στην αρχή η θέση των κρατών μελών δεν ήταν η οριστική τους θέση. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά, ετέθησαν οι πρώτες ερωτήσεις, αλλά ο στόχος μας ως Προεδρία ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το πώς λειτουργεί το σύστημα, τι σχέσεις υπάρχουν μεταξύ ε, των συστημάτων αυτών και τις διάφορες πλατφόρμες ε, για την διαδικτυακή ε, επίλυση διαφορών αλλά και για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και να δουν πόσο ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό και να μπορέσει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ε, και για τα δύο νομοθετήματα. Οι πρώτες αντιδράσεις που είχαμε από αυτές τις συνεδριάσεις είναι οι εξής. Mm, Υπήρξε ένα θετικό μήνυμα από πλευράς κρατών μελών, ε, δεν υπήρχαν αντίθετες απόψεις. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην ε, μελλοντική εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Βεβαίω υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε και τα δύο ε, σχέδια αυτά είναι καινούρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε τα θέματα αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Όσον αφορά τώρα τα ουσιαστικά ζητήματα, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και εδώ στην αίθουσα και αφορούν ε, τις προθεσμίες και για τους δύο κανονισμούς, ε, πότε θα γίνονται ε, οι συναλλαγές και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών και την εισαγωγή αυτών των κανονισμών και φυσικά και τις σχέσεις με το ε, σύστημα με την εναλλακτική επίλυση διαφορών που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Τα θέματα αυτά Συζητήθηκαν στις μέρες αυτές εργασίας στο Συμβούλιο, συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ εναλλακτικού συστήματος επίλυσης διαφορών και του διαδικτυακού συστήματος επίλυσης διαφορών, τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς θα πρέπει να υπάρχει και κάποια επιβάρυνση για τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό που έχει σημασία ε, είναι να δούνε ε, τι ακριβώς ε, θα σημαίνει αυτή η επιβάρηση και τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ότι πρόκειται για ουσιώδη ζητήματα τα οποία ανακύπτουν συνεχώς στη συζήτηση στο Συμβούλιο. Από πλευράς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή σας ε, για τα όσα έκαναν για την προετοιμασία και των δύο νομοθετημάτων και θα ήθελα επίσης να πω και στους συναδέλφους από την ε, μελλοντική Προεδρία και ίσως και την Κυπριακή Προεδρία ανάλογα με την ταχύτητα των εργασιών ε, ότι θα ε, τους εύχομαι και τον δύο ε, να είναι καρποφόρο το έργο τους και να περατωθούν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Et merci aussi... Euh, ευχαριστώ και όλα όσα κάνατε αλλά επίσης υπογραμμίσατε και την τόλμη της Κομισιόν σε σχέση με τον κανονισμό. Και επειδή είναι το τέλος του έτους, θα θεωρώ ότι με μεγάλη ευχαρίστηση εκφράζουμε την ικανοποίησή μας ε, για την επιτυχία αυτή. Και βεβαίως, επειδή οι λεπτομέρειες δεν ξεφεύγουν ποτέ από ε, τις ε, γυναίκες, θα δώσω στις γυναίκες στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο τώρα για να συμπληρώσουν τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει ίσως να καταστήσω σαφές ότι έχουμε και άνδρες συναδέλφους που ήταν που, που ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός στην εκπόνηση του σχεδίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα αξιότιμα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση τα σημεία τα οποία εντοπίσατε φυσικά απαιτούν περισσότερη συζήτηση και διαλεύκανση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα κύρια σημεία χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες και τεχνική συζήτηση. Πρώτον, η διαβούλευση. Με χαρά μπορώ να πω ότι αυτή η διαβούλευση έγινε σε 22 χώρες, ε, γλώσσες, συγγνώμη. 22 γλώσσες. Μία λύπη δηλαδή. Όχι, σε όλες τις γλώσσες της κοινότητας. Είχαμε τώρα έξι συγκεκριμένες απαντήσεις. 32 απαντήσεις από ενώσεις καταναλωτών. Η μεγαλύτερη ομάδα ήταν των επιχειρήσεων, 94 επιχειρήσεις. Και η ανάγκη να κινητοποιηθεί η υποστήριξη από πλευράς επιχειρήσεων πράγματι είναι ε, σημαντική. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν υπέρ της ανάπτυξης συστήματος εναλλακτική επίλυσης διαφορών. Και όλοι καλωσορίζουν την υιοθέτηση και ο Γενικός Διευθυντής της Business Europe λέει ότι αυτή οι φορείς είναι ε, χρήσιμη και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Άρα, ο επιχειρηματικός κόσμος είναι στο πλευρό μας. Δεν είναι μια πρόταση η οποία φέρνει σε αντιπαράθεση επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ένα άλλο θέμα είναι η σημασία της ενημέρωσης. Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι καταναλωτές ότι έχουν δυνατότητες μέσω αυτής της οδηγίας, ότι αυτή η οδηγία τους προσφέρει δυνατότητες και εναλλακτικέ. Και ασφαλώς πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την ενημέρωση. Αυτά όχι βέβαια στις νομικές προτάσεις, αυτά είναι μέτρα αφού υιοθετηθούν οι προτάσεις και αφού αρχίσουν να λειτουργούν φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ε, επίσης, οι ίδιοι εμπορευμόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους καταναλωτές για το ποιοι φορείς θα είναι υπεύθυνοι για την επίλυση διαφορών. Διότι οι ίδιοι εμπορευόμενοι θα συμμετέχουν και θα κάνουν πλήρη χρήση των συστημάτων αυτών. Θα ενημε... Διότι ο επιχειρηματικός κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα συμμετάσχει. Άρα και θα, θα φέρει και το βάρος ή την υποχρέωση, αν θέλετε, ενημέρωσης του κοινού. Στον κύριο Μέιερ, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε εκεί όπου υπάρχουν όλα τα συστήματα εναλλακτικών, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή διαδικτυακών συστημάτων επίλυσης διαφορών. Αυτά τα οποία λειτουργούν ή τα περισσότερα εξ αυτών ε, σε μεγάλο βαθμό ικανοποιούν τις προδιαγραφές, τις ποιοτικές προδιαγραφές της οδηγίας. Κάποιοι φορείς ίσως χρειάζονται κάποια βελτίωση, αλλά όχι πολύ σημαντική. Εξίσου είναι σημαντική η πρόσβαση προς τη δικαιοσύνη. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα τόσο των εμπορευμένων όσο και των καταναλωτών. Και προσέξαμε πολύ ώστε σε όλες τις φάσεις να υπάρχει ενημερωμένη συνένεση εκ μέρους των καταναλωτών να κάνουν χρήση των ADR ή ODR. Και σε περίπτωση μη επίλυσης να μπορούν πάντα να έχουν το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια. Το σχόλιο του κυρίου Ρέπο για την προσπελασιμότητα. Ε, το να έχουν οι καταναλωτές τη μητρική τους γλώσσα όλες τις πληροφορίες. Βεβαίως θα πρέπει αυτή η ανάγκη να ληφθεί υπόψη όταν θα σχεδιάζεται η πλατφόρμα, αλλά η πρόθεσή μας είναι αυτή. Οι καταναλωτές να μπορούν να λειτουργούν στην μητρική τους γλώσσα. Και θα υπάρχουν διευκολυντές διαδικτυακής επίλυσης διαφορών για να υποστηρίξουν τους καταναλωτές στη δική τους μητρική γλώσσα. Αυτό δηλαδή θα περιέχεται στην πλατφόρμα του ODR. Δηλαδή να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ ενός καταναλωτή από μία χώρα μέλος και ενός ε, εμπόρου ή επιχειρηματία που θα βρίσκεται σε άλλη χώρα μέλος. Ένα άλλο θέμα ήταν οι αρχές ποιότητας. Με χαρά εξετάζουμε τις αρχές ποιότητας και ελέγχουμε για την ορθότητά τους. Ε, βασιστήκαμε στις συστάσεις αλλά σίγουρα υπάρχει πεδίο βελτίωσης. Η χρηματοδότηση θα είναι ένα κυρίαρχο θέμα στη συζήτηση αυτή. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ήδη μας ζήτησε να, να, να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησης και να περιληφθεί αυτό στην ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων. και σίγουρα θα χρησιμοποιήσω τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν σε αυτή την Επιτροπή. Και ένα άλλο θέμα είναι η επιτήρηση και οι κυρώσει. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα βαθμό επιτήρηση και εποπτεία. Οι χώρε μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνε ε, ώστε τα συστήματα εναλλακτική επίλυση διαφορών να λειτουργούν σύμφωνα με τι καθιερωμένε αρχέ. Οι κυρώσει που προβλέπονται είναι πολύ περιορισμένε Στην περίπτωση που δεν, ε, που υπάρχει άρνηση παροχής ε, ενημέρωσης και νομίζω ότι θα είναι παρόμοιες οι κυρώσεις με αυτές που προβλέπονται στην ε, οδηγία περί των καταναλωτών, περί των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επίσης, προβλέπονται κυρώσεις και για τα φορείς ε, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που δεν επιτυχάνουν να συμμορφωθούν με τους όρους της οδηγίας. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Είμαι βέβαιη ότι θα υπάρχει πολλή συζήτηση τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το χρόνο που μου διέθεσε. Να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία που αφιέρωσε ήδη τόσο πολύ χρόνο στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή στις συζητήσεις του Συμβουλίου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια δύσκολα ζητήματα που πιστεύω ότι θα επιληθούν τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο, ο οποίος επανήλθε, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το προσωρινό χρονοδιάγραμμα. 24η Ιανουαρίου συνεδρίαση συντονιστών είναι ένα σφιχτό πρόγραμμα, ίσως υπερβολικά σφιχτό. Η προθεσμία για την αποστολή του σχεδίου γρομοδότησης 3 Φεβρουαρίου η εξέταση της νομοδότησης ε, είναι πολύ νωρίς. Κάποιος χωρίς μικρόφωνο. Non, le calendrier a Α, άλλαξε το πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα είναι λιγότερο σφιχτό. Λοιπόν, ακρόαση ανταλλαγή πληροφοριών 29 Φεβρουαρίου, προθεσμία για αποστολή στη μετάφραση στις 4 Μαρτίου, εξέταση του σχεδίου γρομοδότησης στην ΙΜΚΟ 21 Μαρτίου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 30 Μαρτίου 12 το μεσημέρι, εξέταση τροπολογιών 24 ή 27 26 διορθώνει ομιλήτρια. Ε, η ψηφοφορία στις 30 Μαρτίου και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο του 12 που αντιστοιχεί λίγο πολύ στο χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο κύριος Σουάμπ, δηλαδή υιοθέτησε πριν από το καλοκαίρι. Ε, θα δώσω το λόγο στον ε, Πρόεδρο, αφού ευχαριστήσω όλους τους μετέχοντες, την Πολωνική Προεδρία αλλά και την Κομισιόν και το έργο των γυναικών, αλλά επίσης ευχαριστώ και τους άνδρες που συμμετείχαν και που συνεργάστηκαν αρμονικά με τις κυρίες. Και καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, περνούμε στην επόμενη έκθεση και μετά θα αναλάβει ο Μάλκομ. Αλλάζουμε θέμα, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τους πολίτες και τους καταναλωτές. Ερχόμαστε στα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα, συντάξτρια γνωμοδότησης και μετά στους σκιώδεις ε, εισηγητές όσους παρίστανται στην αίθουσα. Κυρία Ιβάνοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα τρόφιμα, για τα βρέφη, τα νεαρά παιδιά και σας παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα να αποχωρήσουν ησύχους, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ιβάνοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθεωρεί τους κανόνες για τρόφιμα που προορίζονται για συγκεκριμένους ε, διατροφικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στην Οδηγία Πλαίσιο 39 του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα νέα κείμενα ε, μετατρέπουν την οδηγία πλαίσιο ε, επιβάλλοντας κάποιους κανόνες για τρόφιμα για αδυνάτισμα, αλλά διατηρώντας και κάποιους κανόνες από το προηγούμενο πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζω την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατηρώντας τις ε, κάθετες οδηγίες για τα βρέφη και τα τρόφιμα για μικρά παιδιά και τα θέματα για τις ειδικού σκοπούς εγκαταλείπεται η έννοια των τροφών για αδυνάτισμα, το οποίο οδήγησε σε κατακαιρματισμό την αγορά και αυτό φυσικά θα μας βοηθήσει να έχουμε υψηλότερο ποσοστό προστασίας για τους ευάλωτες καταναλωτές. Ε, η απλούστευση του υφιστάμενου νομικού πλησίου κατά την άποψή μου θα μειώσει το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα βοηθήσει στην ελεύθερη μετακίνηση αυτών των αγαθών. Η αλλαγή αυτή θα μας βοηθήσει να έχουμε και καινοτομία στον τομέα αυτό, όπου είναι ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς τομείς της ευρωπαϊκής ε, διατροφικής βιομηχανίας. Κάποια βασικά θέματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω τώρα αφορούν ε, τα θέματα ε, για τη γλουτένη. η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την αλλαγή ε, και τα, για τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκι και να περάσουν στον γενικό κανονισμό για τις ε, ισχυρισμούς για τη διατροφή. Θεωρώ ότι θα πρέπει η κατηγορία αυτή τροφίμων να βρίσκεται στο νέο κανονισμό για τις πληροφορίες για τους καταναλωτές και να ισχύουν και οι φυστάμενοι κανόνες για τη σύνθεση και την επισήμανση των προϊόντων και να υπάρχουν ε, οι ίδιες ε, προδιαγραφές προστασίας για την υγεία όπως και σήμερα. Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για τα μικρά παιδιά, τα λεγόμενα γάλατα που βοηθούν την ανάπτυξη και βοηθούν τα νέα παιδιά ηλικία ενό έω τρει έτου και αποτελούν ε, μια ολοένα και αυξανόμενη αγορά σε πολλά κράτη-μέλη. Μέχρι ε, σήμερα δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τα προϊόντα αυτά. Υποστηρίζω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της να ρυθμίζονται τα γάλατα αυτά βάσει ε, του κανονισμού για τη διατροφή και τους ισχυρισμούς για τη διατροφή, για την υγεία, συγγνώμη, και ε, θα θέλαμε να υπάρχουν και ειδικοί κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση και την επισήμανση αυτών των μορφών γάλακτος. Ε, νομίζω ότι αυτό θα αυξήσουν ε, σε μεγάλο βαθμό την προστασία των καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα τις άλλες κατηγορίες ε, των λεγόμενων τροφίμων για αδυνάτισμα, τα οποία είναι εκτός πεδίου εφαρμογή της ε, πρότασης οδηγίας, τρόφιμα για αθλητές, τρόφιμα για αδυνάτισμα και για δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας. Ε, θα θέλαμε οι κατηγορίες αυτές τρομήνων να μπουν στο κανονισμό για τη διατροφή και τους ισχυρισμούς για την υγεία, διότι θα αυξήσουν πολύ περισσότερο τον έλεγχο και την προστασία των καταναλωτών. Για τα τρόφιμα για το αδενάτισμα υποστηρίζω την πρόταση να μπουν στον κανονισμό για τους ισχυρισμούς για τη διατροφή, για τις πολύ χαμηλές σε θερμιδική αξία δίαιτες. Είναι ένα καθόδε ζήτημα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύνθεση την επισήμανση και τη χρήση αυτών των λεγόμενων ε, τροφίμων πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας ε, και ε, έχουμε σύνθεση κάτω από 800 θερμίδες και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται μόνο βάσει ιατρικής εποπτείας, επομένως θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση βάσει της οδηγίας 21 του 99 για τα τρόφιμα για δυνάτισμα για ειδικού ιατρικούς σκοπούς και επίσης προτείνω να υπάρχει και μια ρήτρα opt-out για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν να δεκτούν αυτά τα προϊόντα στην αγορά τους. Επίσης, ε, αναφέρομαι λίγο στη γνωμοδότησή μου και στα θέματα της καινοτομίας, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, τεχνικές και επιστημονικές προόδους που έχουμε, ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιταχύνει τις πράξεις κατεξουσιοδότηση που εγκρίθηκαν βάσει αυτού του κανονισμού για να υπάρξει καινοτομία στον τομέα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω ότι είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία στη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της ε, γνωμοδότησης και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία που έκανε εξαιρετικά ε, καλά τη δουλειά της και φυσικά και όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, οι οποίοι συνεργάστηκαν ιδιαίτερα μαζί μου και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τις απόψεις σας για αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Merci. Donc je donne la parole au... Δίνω το λόγο στους Κιώδης. Στην κυρία Σελά, Σενάλοβα, καταρχήν. Οι άλλοι λάμπουν δια της απουσίας τους αλλά όποιος θέλει μπορεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα των τροφίμων ε, για τις, ε, ε, σε περίπτωση θυλασμού και για, τις, για βρέφη και για ειδικού ιατρικούς σκοπούς θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πιο ευάλωτες ε, κατηγορίες, δηλαδή τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας αυτής της κατηγορίας καταναλωτών. Και νομίζω ότι τα ε, συμφέροντα, κοινοτικά συμφέροντα είναι δευτερεύουσα σημασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πρότασή Υπάρχουν σημεία τα οποία θα συζητήσουμε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων μέσα στα πλαίσια των δικών μας αρμοδιοτήτων. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο τα κράτη-μέλη πρέπει να κοινοποιούν τα τρόφιμα αυτά πριν μπουν στην αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται. Και αυτά τα κριτήρια πρέπει να γνωστοποιούνται για να δούμε κατά πόσο υφίστανται κίνδυνοι για τους καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και εποπτικοί μηχανισμοί. Οι ε, έλεγχοι μετά τη θέση σε εμπορία δεν ε, αρκούν δεν μπορούμε να προβάλλουμε επικίνδυνα τρόφιμα για τα μικρά παιδιά. Στο άρθρο 10 ορίζουμε κριτήρια πληροφόρησης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ε, διάδοση και διαφήμιση στοιχείων από πλευράς επιχειρήσεων. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια επί του θέματος. Υπάρχουν ε, άλλοι ομιλητές επί του θέματος. Ο Αντώνιο. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι σκιώδης σε αυτή την επιτροπή, αλλά σε άλλη. Και γι' αυτό θα ήθελα να παρέμβω και εγώ υποστηρίζοντας ε, τις ε, προτάσεις της εισηγήτριας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία νομοθεσία η οποία είναι αρκετά γενική, οριζόντια δηλαδή, αλλά και εγκάρσια. Νομίζω λοιπόν ότι τα ε, τρόφιμα αδυνατίσματος την χάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης ανάλογα με τη χώρα. Υπάρχει όμως και ένα επίπεδο λεπτομερίας, διότι πρέπει να νομοθετήσουμε, νομοθετούμε και εμείς τομεακά. Η εξαφάνιση της έννοιας τρόφιμα αδυνατίσματος είναι κάτι το ευπρόσδεκτο, καθώς και οι διατάξεις που ε, περιορίζουν τις κατηγορίες τροφίμων που είναι αναγκαίες για ορισμένες ευάλωτες ε, κατηγορίες, όπως τα βρέφη ή προϊόντα με βάση δημιετριακά, προϊόντα για βρέφη και υποπροϊόντα γάλακτος που υποκαθιστούν το θυλασμό. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν και οι βιταμίνες και τα ίχνοστοιχεία που θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Δεν μιλάμε για μια πρόταση που προστατεύει απλώς τον καταναλωτή, έχει και στοιχεία επιστημονικής υφής. Τέλος, Υπάρχει και η υποχρέωση προστασίας της υγείας καθώς και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας διαβούλευσης με την ΕΦΣΑ, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Η προσέγγιση της εισηγήτριας είναι σωστή κατά την απόψή μας, δηλαδή εμβαθύνει τις έννοιες και τα δεδομένα της ε, Κομισιόν και γι' αυτό ε, την υποστηρίζουμε ως πρόταση. Merci. Σας ευχαριστώ πολύ και η συγγήτρια και ο Αντώνιο τόνισαν κάτι πολύ σημαντικό, τα τρόφιμα αδυνατίσματος που διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τα ήθη. Εδώ μιλάμε όχι μόνο για την προστασία καταναλωτών, αλλά και για το σύστημα υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα βασικά στοιχεία και κυρίως επιστημονικά στα οποία αναφέρθηκε ο Αντώνιο. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν κανένας άλλος δεν ζητάει το λόγο. Από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ο κύριος Μαθιουδάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για την έκθεση αυτή. Όπως είπε, Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι η παρέμβασή της καθώς και η παρεμβάση των άλλων ομιλητών διευκολύνει το έργο μας. Γιατί υπάρχει υποστήριξη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Σχετίζονται με προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα γλουτένης ή χωρίς ε, καθόλου γλουτένη. Το επίπεδο προστασίας θα παραμείνει ως έχει γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με κανόνες που έχουν σχέση, σχετίζονται με τη σήμανση αυτών των προϊόντων και άρα τις, ε, οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν σήμερα θα μεταφερθούν στους ε, κατάλληλους κανονισμούς. Η Επιτροπή είχε προτείνει να περάσουν στις αξιώσεις γιατί δεν είχε ε, ακόμα εγκριθεί η οδηγία για την προστασία των καταναλωτών και είχαμε λάβει υπόψη τις υποδείξεις της κυρίας Ιβάνοβα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 36 για πληροφόρηση για τα τρόφιμα προς τους καταναλωτές. Αυτή είναι η κατεύθυνση πολλών μελών του Συμβουλίου. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Σοβαρά εδώ στην Επιτροπή. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα, αλλά προς τα εκεί ρέπουμε. Τώρα πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχουν ορισμένα θεσμικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν γιατί η πληροφόρηση περί τροφίμων στους καταναλωτές ε, αναθέτει, ε, οδηγεί σε κατεξιοδότηση πράξης από πλευράς κομισιών και άρα μπορούμε να υποστηρίξουμε όσον αφορά τις χαμηλές ε, θερμίδες, ε, στα χαμηλά σε θερμίδες τρόφιμα. Δεν υπάρχει ρυθμίση εδώ. Κατανοούμε ότι πολλά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θέλουν να ρυθμιστούν αυτά τα προϊόντα. Μπορώ να πω σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις προτάσεις αυτές εκ του σύνεγγης. Όσον αφορά το ε, γάλα για τα βρέφη, κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια των ε, αξιώσεων. Ως προς την έκθεση Ιβάνοβα, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα λάβουμε υπόψη τις υποδείξεις της. Έγινε μνήα και στις διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, την ΕΦΣΑ. Σας είπα ότι για λόγους δημόσιας υγείας, όταν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, πάντα ε, γίνονται διαβουλεύσεις με την ΕΦΣΑ και υπάρχει και η πρόταση Υπάρχει μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαι σίγουρος ε, κατά πόσο κατανόησα την παρέμβαση για τις ε, κοινοποίησεις οι κοινοποίησεις προβλέπονται στους ειδικού κανόνες για τα τρόφιμα, για ιατρικούς σκοπούς. Άρα θα κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα στους ειδικού κανόνες. Εδώ μιλάμε για τη γενική πλαισίωση και ως προς τις ως προς τα καινοτόμα στοιχεία, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι κανονισμοί έτσι ώστε να συμβαδίζουν με την τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν άλλα σημεία και νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα, στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν, αλλά και την Επιτροπή για τα σχόλιά της. Σημείωσα τα σχόλιά σας. Κυρία Σινιαλόβα, υποστηρίζω αυτό που είπατε, δηλαδή την ανάγκη αύξησης των μηχανισμών ελέγχου. Γι' αυτό προτείνω ένα νέο εδάφιο το 27Γ που ζητά από τις χώρες μέλη να διεξαγάγουν ελέγχους για την συμμόρφωση προς τον κανονισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο, με το οποίο συμφωνεί ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ασφαλώς συμφωνώ ότι χρειάζονται περισσότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί Έχουμε βεβαίω τον κανονισμό, αλλά ποιο συμμορφώνεται και ποιο όχι είναι διαφορετικό θέμα. Γι' αυτό επιμένω στο να υπάρξει και αυτό το εδάφιο το 27 γ Πέραν τούτου δεν έχω πολλά να προσθέσω. Σας ευχαριστώ όλους για μία ακόμα φορά. Και σας εύχομαι καλές γιορτές. Euh, ε, ευχαριστώ. Η... η Πολωνική Προεδρία απεχώρησε. Πιστεύω ότι θα παρέμβει στις επόμενες. Τώρα, προσωρινό χρονοδιάγραμμα. Εξέταση, η, μάλλον η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 12 Ιανουαρίου. Εξέταση τροπολογιών 6 Φεβρουαρίου. Α, να τελειώσω το χρονοδιάγραμμα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα αν θέλει να εκφραστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει εξέταση τροπολογιών 6 Φεβρουαρίου. Ε, την ίδια μέρα όμως έχουμε και την ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ. Ε, πώς θα γίνει αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Mm. Oui, θα δούμε αν αυτό είναι δυνατό, διότι υπάρχει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η ψηφοφορία στις 29 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο του 12. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά αν έχουμε και άλλες συνεδριάσεις. Εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε στις αρχές του Ιανουαρίου. Κυρία Παρβάνοβα, επειδή είστε ε, σκιώδης ε, εισηγήτρια από την άλλη, δεν θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Ε, είστε πολύ ευγενικοί. Σήμερα ήταν μια τρελή ημέρα. Τρέχουμε δεξιά-αριστερά. Uh, uh, uh, πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα Άλντε καλωσορίζει την πρόταση αυτή στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ε, που ήταν απαραίτητη για την προστασία των καταναλωτών. Χρειάζεται πράγματι ειδική νομοθεσία για τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο για τις ευάλωτες ομάδες. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ιβάνοβα για το σχέδιο που παρουσίασε και εξ ονόματος της ομάδας μου μπορώ να πω ότι υποστηρίζουμε την προσέγγιση που υιοθέτησε η κυρία Ιβάνοβα. Πολύ σύντομα θα παρουσιάσω κάποια σημεία. Πιστεύω ότι η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα τα επεξεργαστεί περαιτέρω. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή είχε τη συζήτηση της... Ε, ε, συζήτησε μάλλον το σχέδιο και γίνεται η πρόταση τα τρόφιμα τα οποία ε, έχουν να κάνουν με ειδική ενεργειακή διατροφή ή ειδική διατροφή θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής νομοθεσίας. Και ως προς το ε, σκέλος των τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά. Συμφωνώ με την κυρία Ιβάνοβα και με την πρόταση της Κομισιόν ότι αυτά θα πρέπει να είναι πάντοτε κάτω από την νομοθεσία σχετικά με την προστασία της υγείας και του καταναλωτή. Και ασφαλώς πρέπει να, υπάρχουν και, να υπάρχει κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση. Ε, Επίσης, ε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ορισμοί σχετικά με τη σύνθεση των βρεφικών ε, τροφών και των τροφών για μικρά παιδιά και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο βασικό νομοθετικό κείμενο και να ακολουθηθεί η κανονική νομοθετική διαδικασία. Και ως προς την προληπτική αρχή, αυτή θα πρέπει να είναι μια κεντρική αρχή κανένα τρόφιμο δεν θα πρέπει να τίθεται στην αγορά αν θεωρείται ύποπτο ή επικίνδυνο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των ε, πολιτών που καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί ως προς την ε, παρουσία στις τροφές αυτές ε, ε, ζυζανιοκτώνων και άλλων ε, ουσιών. Αυτά είχα να πω και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση από όλους. Η, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η συγγήτρια δεν θέλει να λάβει το λόγο. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε ακριβώς την ώρα μας στο επόμενο θέμα και δίνω αμέσως το λόγο στον Πρόεδρό μας. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε την ομάδα που ασχολείται με τα τρόφιμα να αποχωρήσει από την αίθουσα, διότι είναι ευαίσθητη τους θορύβους. Έχουμε όμως και την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση IT. Να καλωσορίσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που μας παρουσίασε την αξιολόγηση αντικτύπου πριν από κάποιο καιρό και εργάζεται για το θέμα αυτό. Η κυρία Κόρχολα και εγώ ήμασταν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, νωρίτερα και ήρθαμε απευθεία από εκεί και η κυρία Κόρχολα θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις της τώρα. Χάσαμε τον κύριο Ταραμπέλα, τον καλωσορίζουμε όμως γιατί είναι εδώ σήμερα και δεν είναι μόνο ως ο ε, συζητής εδώ, αλλά ανέλαβε και για το 2012 την έκθεση για την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες. Πάμπολες σελίδε. θα έχετε πολύ ωραίο ανάγνωσμα για τι διακοπέ σα, αλλά θα είναι ζωτική σημασία στο ζήτημα αυτό για μας. Σας καλωσορίζουμε όμως τώρα ως σκιώδη συζητή για την περιαγωγή. Έχουμε... Ε, και άλλους εδώ. Ε, ο κύριος Μπίνιγκεν δεν είναι εδώ. Μπορεί να πω εγώ ένα-δυο πράγματα εξ ονοματός του. Ο κύριος Γκυγιόμ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σλαβίν δεν είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε απαρτία σχεδόν εισηγητών, επομένως ε, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κόρχολα για να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε, με την οποία έχουμε ενισχυμένη συνεργασία για το θέμα αυτό. Ρίτα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Μάλκομ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Όπως θα γνωρίζετε, πρέπει ο κανονισμός για την παραγωγή 3 να ε, ετοιμαστεί σύντομα και να έχουμε και συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση δυνατών, ώστε να μην υπάρχει κενό και να μην υπάρχει ε, κανονισμός για την περιαγωγή ενισχύ. Έχουμε κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή Βιομηχανίας για αρκετά ε, άρθρα και το μόνο άρθρο το οποίο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ε, η Επιτροπή ε, Βιομηχανίας και για την οποία δεν έχω καταθέσει τροπολογία είναι το άρθρο 3 ε, για τη χοντρική πρόσβαση. Δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε τα θέματα αυτά και το ίδιο ισχύει και για τα ανώτατα όρια για τη λιανική και χοντρική πώληση. Επομένως η ΙΤΡΕ και η Επιτροπή μας θα ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Η Επιτροπή Βιομηχανίας βέβαια έχει και το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών που καλύπτονται αρκετά καλά στην πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δούμε τις επιπτώσεις της τρέχουσας νομοθεσίας για την περιαγωγή από το 2007, η οποία τροποποιήθηκε το 2009, διαπιστώνουμε ότι μείωσε ουσιαστικά την τιμή και των κλήσεων αλλά και των μηνυμάτων ε, περιαγωγής, αλλά... Ε, οι περισσότερε τιμέ είναι κοντά στα ανώτατα όρια που ε, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει ο κατάλληλο ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους στόχους της για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα δήλωσε ότι οι τιμές και οι διαφορές στην περιαγωγή θα πρέπει να φτάνουν στο 0 ε, μέχρι το 2015 και για να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο αυτό θα πρέπει να έχουμε μια λύση η οποία θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς περιαγωγής και μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Να πω και ένα-δυο λόγια για τα διαρθρωτικά μέτρα και τα ανώτατα όρια τιμών. Συζητάμε αρκετές διαδοτικές αλλαγές ε, πιο ε, αναλυτικά, το dual MC, το local breakout και όλα αυτά, τα οποία όλα έχουν και πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και πολλά μειονεκτήματα και βεβαιότητε. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πολύ νωρί για να καθορίσουμε ποια θα είναι η καλύτερη λύση μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό ε, θα ήταν και γελίο να ε, νομοθετήσουμε για την τεχνική λύση που θα πρέπει να επιλέξουμε, διότι μπορεί να δημιουργήσουμε νομοθεσία η οποία να είναι ήδη ε, παροχημένη όταν θα τεθεί σε εφαρμογή. Η τεχνολογία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, γι' αυτό και επέλεξαν να ε, τροποποιήσω τον κανονισμό αναφέροντας τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει τελική τεχνική λύση. Όσον αφορά τώρα τα ανώτατα όρια, πρότεινα κάποιες αλλαγέ και θα καταθέσουμε και κάποιες άλλες αλλαγέ αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει αρχικό περιθώριο μεταξύ ε, τιμών χονδρικής και τιμών λαϊλιανική και να είναι 2,4 με 3 φορές ε, περισσότερες ε, από την ε, χονδρική πώληση τιμές της Λιανικής, ώστε να υπάρχει και ένα λογικό κέρδος και τα ανώτατα όρια να μπορέσουν να ε, αρθούν στο μέλλον. Όλοι θεωρούμε ότι οι παρούσε τιμέ είναι γελίε, αλλά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καλά λειτουργούσα αγορά για τις τιμές περιεγωγές, θα πρέπει να υπάρχουν ανώτατα όρια σε λογικό επίπεδο για να προσελκύσουμε και νέου επενδυτέ για να έχουμε και τον κατάλληλο ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τα ανώτατα όρια μετά από το 2016, διότι υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί χρόνος για να αναπτυχθεί αγορά. Δεν έχω αλλάξει τις προθεσμίες προς το παρόν, αλλά θα θέλαμε να τις αλλάξουμε αργότερα εντό του μηνός. Όσον αφορά τώρα την προστασία των καταναλωτών και τη διαφάνεια, ε, η διαφάνεια στις τιμές βελτιώθηκε σημαντικά με τη θέσπιση των προηγούμενων κανονισμών για την περιογωγή, αλλά αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν. Ε, οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο και να μπορούν να συγκρίνουν και πιο εύκολα τιμές και ενδεχομένως να αλλάζουν και πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής. Με τις τροπολογίες που κατέθεσα προτείνω ε, το όριο ασφαλείας των 50 ευρώ ή ένα ανώτατο όριο το οποίο θα διαμορφώνεται σε προσωπική βάση να επεκταθεί και στο υπεραγωγή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν ειδοποίηση από τον πάροχο όταν πλησιάζουν το όριο ασφαλείας της περιαγωγής τους. Επίσης πρότεινα να επεκταθούν αυτά τα μέτρα και για προπληρωμένες υπηρεσίες, διότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να λάβει κάποιος υπέρογκο λογαριασμό, ακόμα και αν είναι προπληρωμένα τα συμβόλαια. Ε, ως γενική παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι οι πληροφορίες για τους καταναλωτές ε, ελήφθησαν δεόντως υπόψη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να προσπαθήσει να επιτύχει μια σαφέτερη, σαφέστερη δομή του κανονισμού, εξορθολογίζοντας όλες τις διατάξεις που αφορούν ε, την προστασία του καταναλωτή και για τους υπέρογους λογαριασμούς και για τις απαιτήσεις διαφάνειας που αφορούν για όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια. Ε, Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Ας μιλήσουν λοιπόν οι σκιώδεις ο κύριος ε, Ταραμπέλα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τις υποδείξεις σας για να αναγνώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα στο τέλος, της, ε, το νέο, μάλλον στο τέλος του έτους και με τις γιορτές. Έχουμε πολύ ε, διάβασμα γιατί θα ασχοληθούμε και με τον κανονισμό για τις δημόσιες προμήθειες. Μιλάμε για την καταβληθήσα τιμή σε SMS όχι μόνο στη χώρα αλλά και εκτός. Αυτοί που χρησιμοποιούν καρτοκινητή τηλεφωνία θα πρέπει να έχουν τις ίδιες πληροφορίες και την ίδια προστασία με τους υπόλοιπους. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ο στόχος της επικείμενης ρύθμισης με βάση την ψηφιακή ατζέντα της Κομισιόν οδηγεί σε ισότητα τιμών μέχρι το 2015 ως προς τις εσωτερικές επικοινωνίες και την περιαγωγή. Όμως η Επιτροπή δημιουργεί δύο αγορές. Την ε, αγορά των εθνικών τιμών και την αγορά της περιαγωγής. Αυτό είναι επιζήμιο για τους καταναλωτές ως προς την ε, πληροφόρηση. Αν θέλουμε ενιάγορα μέχρι το 2015 θα πρέπει να προτείνουμε ε, πιο ρηξικέλευθες λύσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ανώτατες λιανικές τιμές έτσι ώστε να μειωθούν καταρχήν έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει δελεαστικές τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει οι ανώτατες τιμές θα πρέπει να ισχύσουν μέχρι το 2016. Μέχρι όμως τον Ιούλιο του 2014 οι τιμές περιαγωγής και οι εθνικές τιμές θα πρέπει υποτίθεται να είναι οι ίδιες. Δεν θα πρέπει απ' την άλλη να αυξηθούν οι εθνικές τιμές. Σε ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο που γνωρίζω σχετικά καλά, οι εθνικές τιμές είναι υψηλότερες από τις τιμές περιαγωγής για τα SMS. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι για να μειωθούν οι τιμές της περιαγωγής. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε, να φτάσουμε στην ενιαία αγορά επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας, και θα υποβάλω τροπολογίες έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους ανηλίκους ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό το σοκ των λογαριασμών όπως είπε και η κυρία Κορόλα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τιμολόγηση της τηλεφωνίας και ιδιαίτερα σε σχέση με την περιαγωγή. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης που διέπει την Κομισιόν. Δεν με δελεάζει η ιδέα να ε, μειωθούν οι τιμές με εικονικούς παρόχους. Ο καθένας ξέρει το επάγγελμά του. Οι πάροχοι ξέρουν τη δική τους. Θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές, αλλά δεν θα ήταν σκόπιμο οι μεγάλες επιφάνειες, ας πούμε, να ασχοληθούν με την περιαγωγή, να αναλάβουν μόνο την ε, περιαγωγή και όλοι οι άλλοι πάροχοι την τηλεφωνία γενικά. Θα πρέπει να αναγνώσουμε την ανακοίνωση, αλλά δεν νομίζω ότι με εικονικούς παρόχους θα μειώσουμε την τιμή της περιαγωγής. Δεν με δελεάζει αυτή η ιδέα και σας το λέω εξ αρχής, δεν θα τη λάβω υπόψη σοβαρά. Πάση περιπτώσει είμαστε στην ε, απαρχή των συζητήσεων. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, η τα τιμολόγια της περιαγωγής δίδουν ε, στον Ευρωπαίο καταναλωτή την ε, γνώση σχετικά με την κινητικότητα στην Ευρώπη. Και η μείωση των ε, τιμών είναι κάτι χαρακτηριστικό. Πολλά από τα σχόλια που έκανε η κυρία Κόμπολα, με πολλά εξ αυτών συμφωνώ. Ε, οι τιμές που καθορίζονται από τους παρόχους ε, μάλλον επιβάλλονται από τους παρόχους και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ε, μείωση, η περικοπή αυτών των τιμών. Αυτή τη στιγμή η αγορά ελέγχεται από ολιγοπόλια. Αυτό όμως θα πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι θα, είναι, θα δέχονται μία τιμή η οποία θα είναι ενδιαφέρουσα και για αυτούς και για την αγορά. Αυτό είναι πολύ απλό για να επιτευχθεί. Ωστόσο, αν πάμε σε πολύ χαμηλές τιμές, δεν θα υπάρξουν νέοι πάροχοι. Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή. Από την άλλη, αν οι τιμές πάνε πολύ ψηλά, τότε οι κατανοητές δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Διότι οι κατανοητές είναι αυτοί που πληρώνουν τις υψηλές τιμές ε, περιαγωγής. Η Κομισιόν ε, κάνει μνήα σε μια ευρεία ρύθμιση της αγοράς στο μέλλον. Δεύτερο σχόλιο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ή να σκεφτούμε νέες τρόπους, νέες μεθόδους και νέες τεχνικές ώστε να υπάρχουν ενιαία δίκτυα ή υπερεθνικά δίκτυα ώστε να μην χρειάζεται η περιαγωγή. Η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, εξετάζει μια ενιαία τιμή ώστε ο εθνικός ε, πάροχος να δηλώνει ότι έχω μια ενιαία τιμή για την ε, περιαγωγή. Αυτό το οποίο Ε, επιβαρύνεται ας πούμε στην συνομιλία ή στα SMS είναι ακριβώς τα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται. Αυτά είναι και τα πακέτα δεδομένων τα οποία προκαλούν αυτό που αποκαλείται σοκ λογαριασμών. Αν λοιπόν έχουμε και μία λογική τιμή για τα πακέτα δεδομένων, τότε θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα εφαρμογής, τα οποία θα πρέπει και αυτά να τα εξετάσουμε. Αν είμαι τώρα ένας τακτικός χρήστης, τότε θα πρέπει να σκεφτώ μια εναλλακτική λύση. Για να μπω κατευθείαν στο δίκτυο δεδομένων, στο τοπικό δίκτυο δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα τα δεδομένα και τις τεχνικές πτυχές. Η βεβαίως τεχνολογική πρόοδος είναι ραγδαία. Πρέπει να σκεφτούμε και τις εναλλακτικέ αυτών που προτείνει η Κομισιόν. Το θέμα δεν είναι απλό, αλλά νομίζω ότι αξίζει προσπάθεια. Αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι εναλλακτικέ θα είναι φθηνότερες ακριβές επενδύσεις μπορεί να μην αποδίδουν υπέρ του καταναλωτή και υπέρ των χαμηλών τεχνολογιών. Πρέπει λοιπόν από κοινού να σκεφτούμε εάν υπάρχουν εναλλακτικέ στις προτάσεις της Κομισιόν, οι οποίες όμως θα είναι υπέρ και προς το συμφέρον του καταναλωτή, διότι αυτό είναι το νόημα. Πώς μπορούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω την εσωτερική αγορά και να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ο καταναλωτής θα έχει φθηνότερη τηλεφωνία καθώς κινείται εντός της Ευρώπης. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Η Κομισιόν κάνει αυτές τις γενναιόδορες προτάσεις για την είσοδο στην αγορά εκεί όπου δεν υπάρχουν υποδομές. Αυτό είναι καλή ιδέα καταρχήν, αλλά ακούω ότι υπάρχει ε, ε, διατυπώνονται ιδέες για μείωση αυτών των δυνατοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι αρκετά ελκυστική πλέον η αγορά για νέους εισερχόμενους. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού είναι το κλειδί για φθηνά τιμολόγια. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τις προτάσεις της κυρίας ε, Κόρολα και τις εναλλακτικές που υπάρχουν σε ένα σχέδιο οδηγίας βεβαίως μπορεί κανείς να περιλάβει όλες τις εναλλακτικέ και να αφήσει την αγορά να αποφασίσει και να επιλέξει και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το καλύτερο για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κρίστιαν Ένστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι ένα από τα θέματα που αγαπώ διότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι που είναι πολύ καλό για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα είναι υπέρ και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όταν ε, είσαι ας πούμε επιχειρηματίας ε, και ε, επισκέπτεσαι διάφορες χώρες μέλη, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου με σε λογικές τιμές και οι περιορισμοί που υπήρχαν στην περιαγωγή ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο. Πολλά όμως ρυθμίζονται αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της υπερβορικής ρύθμισης, όχι παραπάνω από ότι είναι οι υπόλοιποι παρόντες στην αίθουσα αυτή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητη, διότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών δεν είναι απλώς ένας κλάδος. Είναι ο βασικός κλάδος που βοηθάει όλους τους υπολείπους. Δεν μπορεί κανένας να δουλέψει χωρίς τηλέφωνο στις μέρες μας. Συμφωνώ λοιπόν με τα γενικά σχόλια. Πρέπει να μπει κάποια τάξη και συμφωνώ και με τα ε, γενικότερα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με την προστασία των καταναλωτών έναντι των σοκ των λογαριασμών, ακόμα και όταν πρόκειται για ε, κλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Σήμερα στην ακρόαση η κυρία Νίμπελ έλεγε, αναφερόμενη στην Deutsche Telekom, η Κάζο, ότι προσφέρουν το τοπικά πακέτα για 8 GB ενώ ε, στην Ισπανία ε, προσφέρουν για 2 GB, 2 GB για 12,5 ευρώ το μήνα. Στη Σουηδία οι τιμές λίγο πολύ είναι ίδιες, αλλά τούτο μας δείχνει και το μέγεθος Πιστεύω λοιπόν ότι ε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μείωση τιμών, δηλαδή ένα σέντ ένα 10 ευρώ το gigabyte ας πούμε χοντρικά και αυτό δίνει πολύ περιθώριο και για κέρδος για τους ε, ε, για τις εταιρείε. Ε, βεβαίως, η τιμή της χονδρικής είναι η καθοριστική που θα επιτρέψει και στους, ε, στις εταιρείες να μπουν κανονικά στον ανταγωνισμό και να μπορέσουν να λειτουργήσουν υπέρ των καταναλωτών. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Κρίστιαν, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες. Και ο κύριος Μπίλαν έστειλε κάποια σχόλια, κάποιες σημειώσεις, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Γενικά υποστηρίζει την γενική προσέγγιση της κυρίας ε, Κόρολα. Και νομίζω ότι συμμερίζονται την άποψη αυτή και τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας. Πρέπει να υπάρξουν δηλαδή κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές για να επιταχυνθεί ο ανταγωνισμός και να εισαχθούν νέοι τρόποι ε, παροχής δυνατοτήτων επιλογής από τους καταναλωτές. Και πιστεύω ότι αυτή η άποψη διατυπώθηκε και από τον ε, Μπέρεκ Νομίζω ότι ήταν στη δεύτερη συζήτηση αυτού του φακέλου. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Jim Nimblitz στην Επιτροπή που ε, είναι σύμβουλο σχετικά με θέματα κανονισμού περιαγωγής. Θεωρώ ότι είναι ένας βετεράνος αυτής της διαδικασίας, διότι έχει συνεισφέρει πολλά Νομίζω ότι η γενικότερη κατεύθυνση που προτείνεται τόσο από, από αμφότερους τους, στρατη, τους είναι αντιληπτή. Χρειάζεται να υπάρξει ένα καθεστώς ε, ορίων ε, τιμών για να προχωρήσει η αγορά, να μειωθούν τα κόστη και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και όπως ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι, το θέμα καθορισμού των τιμών χονδρικής ε, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων και ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό σύστημα περιαγωγής αγοράζοντας χρόνο ή λεπτά ή ε, gigabytes από άλλους παρόχους για να προσφέρουν κάλυψη σε ολόκληρη την Ένωση. Άρα λοιπόν το όλο θέμα της χονδρικής τιμής είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως είπε και ο Κρίστιαν. Από την άλλη πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν θέλουμε μια μόνιμη λύση αυτό θα απαιτήσει διαρθρωτικές αλλαγές Δηλαδή πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και πρέπει να υπάρξει απόδοση αυτών των επενδύσεων. Ο Κρίσιο νομίζω έχει δίκιο όταν ε, μιλάει για μείωση των τιμών στα μεταφορά δεδομένων, αλλά η κατανάλωση των δεδομένων συνδέεται πολύ περισσότερο με την τιμή από ότι ας πούμε η, τα, η φωνητική τηλεφωνία. Μπορούμε δηλαδή να, έχουμε ένα νέο σύστημα τιμών και αυτή τη στιγμή οι ε, πάροχοι να επενδύουν σε περισσότερο, ε, σε μεγαλύτερες χωρητικότητες, μεγαλύτερο όγκο. Από την άλλη μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση και να μην υπάρχει επαρκής ε, διαθέσιμη χωρητικότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμό. Χρειάζεται να επενδύσουν επίσης στις νέες σε, σε, τεχνολογίες νέας γενιάς με μεγαλύτερες χωρητικότητες. Επίσης υπάρχουν ε, αυτά τα νέα συστήματα ευρυζωνικότητας, οι νέες προτάσεις οικουμενικής ευρυγωνικότητας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις μεμονωμένα χωρίς να λάβουμε υπόψη και ε, την, την διάσταση αυτή της ε, εξέλιξης. Άρα λοιπόν με βάση τις προτάσεις που κάνει η κυρία Κόρολα, δεν, πρέπει να είναι αυτή, αυτό το κείμενο πολύ περιγραφικό και λεπτομερές ως προς την τεχνολογία. Θα πρέπει να προσφέρει λύσεις και βεβαίως το όλο θέμα θα πρέπει να ελέγχεται. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και επαρκής χρόνος ώστε να μπορέσει η αγορά να αντιδράσει κανονικά νέες λύσεις και η, νέα, η εισαγωγή των νέων λύσεων στην αγορά δεν γίνεται πολύ γοργά. Άρα λοιπόν πρέπει να επιτρέψουμε και στην αγορά να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί και να επανέλθουμε. Ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια θέση όπου αυτό το κοινοβούλιο διαρκώς θα πρέπει να ε, θεσπίζει κανονισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πανευρωπαϊκές υπηρεσίες, διότι δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Το κάναμε αυτό επειδή υπήρξε ε, έλλειψη βούλησης ή ανικανότητα από πλευράς ε, παρόχων. Αλλά δεν θέλω να, έχουμε περιαγωγή 3, 4 και 5 στο μέλλον. Αυτά λοιπόν, ε, μίλησε ο κύριος, έχει το λόγο. Συμφωνώ ότι καταρχήν δεν θα πρέπει να ορίσουμε τιμές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο Αγορά θα τις ορίσει. Αλλά δεν εμπιστεύομαι την αγορά αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανταποκριθεί. Γι' αυτό θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Νομίζω ότι η αγορά είχε αρκετό καιρό. Εγώ το 2006 εξελέγην εδώ όταν συζητήσαμε την πρώτη, τον πρώτο κανονισμό περί περιαγωγής και είπαμε ότι χρειάζεται να δώσουμε χρόνο στις αγορές. Τώρα μιλάμε για το 2015, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν οι αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα στεναροί και θα πρέπει κάτι να κάνουμε και με την τιμολόγηση. Δεν συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν, πολύ υψηλές τιμές. Κυρία Κορχόλα, οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Συμφωνώ με τον ε, Κρίστιαν ότι δηλαδή οι τιμές χονδρικής θα ήταν ένα καλό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία τιμολόγηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε χαμηλή τιμή χονδρικής ως τιμή εκκίνησης. Το συζήτησα και με πολλά λόμπι από πλευράς ε, βιομηχανίας. Και μερικοί λένε ότι είναι δυνατόν να έχουμε μία ανώτατη τιμή χονδρικής 10 ευρώ. Και πάλι θα είχαν μεγάλο κέρδος, γιατί Εάν η τιμή είναι χαμηλή, τότε οι καταναλωτές δεν θα φοβούνται και οι επιχειρήσεις δεν θα φοβούνται να χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι τους τα εφή e τηλέφωνα. Άρα δεν θα κερδίζουν ανά γιγαμπάιτ, αλλά από το γεγονός ότι πολλοί θα χρησιμοποιούν e, εφή συστήματα, εφή e προϊόντα. Κάτι έχει γίνει, κάτι ελπίζω ότι θα γίνει κατά τη Δανέζικη Προεδρία και ελπίζω το Κοινοβούλιο να δεχτεί να μειώσουμε τις τιμές και να μην το αφήσουμε στο Συμβούλιο. Δεν μπορεί το Συμβούλιο να υπερασπιστεί τους καταναλωτές. Αν δεν μειώσουμε τις τιμές, τότε το Συμβούλιο θα πει ότι θα πρέπει να έχουμε χαμηλές τιμές εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ΜΜΕ και με τους καταναλωτές. Συμφωνώ με τον Κρίστιαν για την τιμή χονδρικής και με βάση αυτή θα πρέπει να εργαστούμε. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε και για τον τελικό χρήστη βεβαίως. Και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι η δική μας Επιτροπή είναι η Επιτροπή επί της ουσίας και θα πρέπει να μιλήσει για τις καλύτερες ε, τιμές για τους καταναλωτές. Και η πρόταση ε, Κορχόλα είναι υψηλή και πολύ πιο υψηλή από την πρόταση της Ήτρε. Δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε ως προς τις τιμές εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν δυνατότητες για χαμηλές τιμές χονδρικής χωρίς να βλάψουμε τις εταιρείε. Και έτσι θα έχουμε κάνει και κάτι καλό για τους καταναλωτές. Άλλη, η κυρία Τούν. Ευχαριστώ. Θα προτιμούσα οι επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλά τις τιμές να τις ορίσουν καλά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αλλάζουμε πάροχο για την περιαγωγή. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί όλοι όσοι ταξιδεύουν βάζουν την ε, περιαγωγή εκτός. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό για την εσωτερική αγορά, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τιμές, ε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια, να τα ελέγξουμε και γι' αυτό βάζουμε το data roaming off όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Η κυρία Ράτη μας είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τη, τους υπολογιστές όταν είμαστε στο 14ο όροφο. Μα μας είπε, εσείς έχετε τα smartphone σας, άρα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Όμως είναι ένα δαπανηρό εγχείρημα και κάτι θα πρέπει να γίνει. Επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων, θα πρέπει να τις το επιβάλλουμε, τους το επιβάλλουμε ακούγαμε εδώ και πολλά χρόνια ότι θα προπτωχεύσουν αν ε, μειώσουμε τις τιμές. Μα όλο ένα και μειώνονται οι τιμές και κανένας δεν πτωχεύει ίσα ίσα. Λειτουργούν ακόμα καλύτερα και με υψηλότερα κέρδη. Μαθαίνουμε από τις επιχειρήσεις ότι έχουν διαφορετικές τιμές αναχώρα και εξαρτάται από τον πλούτο του πολίτη τι χρήματα μπορεί να καταβάλει, αλλά και στις φτωχές χώρες κερδίζουν αρκετά καλά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Άρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ελιγμού και οι τιμές μπορούν να χαμηλώσουν. Φοβάμαι λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι τάσσομαι κατά της εικόνας αυτής που δημιουργείται για τις αγορές, θα πρέπει να χαμηλώσουμε τις τιμές που θα είναι καλές και για τις επιχειρήσεις, γιατί θα χρησιμοποιούμε περισσότερο το διαδίκτυο, θα είναι πολύ καλό για την εσωτερική αγορά και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Και αυτό θα είναι πολύ καλό και για την ασφάλεια. Κορέια Ντεκάμπος. Ευχαριστώ Μάλκομ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι όλοι παρευρεθήκαμε στην ακρόαση της Επιτροπής Ήτρε όπου μάθαμε ότι οι παρούσες τιμές περιαγωγής αποτελούν πολλαπλάσιο του κόστος. Κάτι μεταξύ 5 και 10, επί 5 ή επί 10. Αυτό σκανδάλισε τους παρόντες και ρωτήσαμε την Επιτροπή γιατί ισχύει κάτι τέτοιο. Και μετά από πρώτη, από την πρώτη μείωση τιμών, γιατί να μην έχουμε και μία δεύτερη. Η Επιτροπή μας είπε ότι οι τιμές είναι αρκετά υψηλές έτσι ώστε να ενισχύσουμε, να ενθαρρύνουμε επιχειρήσεις να μπουν στην αγορά. Μα αυτό είναι αβάσιμο, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σχεδόν, με, ένα ιονί μονοπόλιο, με ένα ε, ολιγοπόλιο, διότι τη στιγμή που ορίζονται ανώτατα όρια, τώρα υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν οι τιμές και μετά προβλήθηκε και ένα άλλο επιχείρημα. Μα ήδη υπάρχει ανταγωνισμός. Ε, δηλαδή, όταν βγαίνουμε από τη χώρα μας, λαμβάνουμε ένα μήνυμα όπου έχουμε την νέα τιμολόγηση, την τιμολόγηση περιαγωγής. Πώς οι καταναλωτές όμως αλλάζουν πάροχο επειδή ακριβώς λαμβάνουν αυτή την ε, πληροφορία. Δηλαδή, το, την κοιτάνε αυτή την πληροφόρηση ή βιάζονται για να πάρουν τη βαλίτσα τους και να φύγουν για την πόλη. Δηλαδή, υπάρχει σωρία επιχειρημάτων που είναι αβάσιμα. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Κορχόλα ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση αλλά ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προτάσεις του Μαρκ Ταραμπέλα. Δηλαδή να υπάρχει ένας μηχανισμός για να φτάσουμε σε ε, ένα νέο φάσμα οροφών μέχρι το 2015. Έτσι θα ωφελήσουμε τους ψηφοφόρους μας. Θυμάμαι ότι μέσα στα πλαίσια των πληροφοριών που μας δίνονται, μία από τις υπηρεσίες είναι η περιαγωγή και είχαμε ένα πρώτο κύμα μειώσεων των τιμών. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε και στο δεύτερο κύμα μειώσεων. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Θα ήθελα η Επιτροπή κάτι να μας πει επί του θέματος. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυρία Νίμπλερ. Ε, έχουμε 7 λεπτά πριν από το κοκτέιλ μας και θα συνοψίσει η κυρία Κορχόλα στο τέλος. Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμένα είναι το αγαπημένο μου θέμα η περιαγωγή, όχι γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή, αλλά για τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Άξτρομ, το πόσο σημαντική είναι η περιαγωγή για την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και να συνεχίσω ε, από αυτά που μόλις άκουσα. Η κυρία Κόρχολα στην παρουσίασή της έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση δηλαδή ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων, διαρθρωτικών μέτρων, για την εισαγωγή ανταγωνισμού στην αγορά και ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα ε, δίκτυο ασφαλείας στους καταναλωτές ε, για τις ανώτατες τιμές και νομίζω ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά τα μέτρα μεταξύ των αν θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό στην αγορά περιαγωγής που νομίζω ότι είναι και ο στόχος για όλους μας. μία επιπλέον παρατήρηση για τα υπεραγωγή δεδομένων, για το data roaming. Όπως είπε και ε, κάποιος, αυτό είναι το μέλλον ε, στην περιαγωγή. Χρησιμοποιούνται υπηρεσίες roaming ε, και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά θα ήθελα να μπορούν να χρησιμοποιούν και το data roaming όταν ταξιδεύουν. Και αυτό που κατέληξε ο συμπέρασμα κυρία Κόλχολα, ναι, είναι λογικό. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες για τις λύσεις, αλλά γνωρίζουμε από τις αναλύσεις ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις διαθέσιμες και θα πρέπει στον κανονισμό να καθορίσουμε τα κριτήρια προκειμένου να επιλέξουμε τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις κατά τρόπον ώστε να μην αποκλείσουμε τις νέες κοινοτόμες λύσεις. Και πιο συγκεκριμένα, ε, λύσεις οι οποίες ε, θα ε, αντιμετωπίζουν τις υψηλές τιμές σε data roaming και τις αυξανόμενες προσφορές στην αγορά των πακέτων δεδομένων. Θα θέλαμε να ρυθμίσουμε τις περιαγωγές πακέτων δεδομένων σε πολύ χαμηλή τιμή, ώστε να μπορούν να έχουν προσιτές τιμές για το data roaming, αλλά ακόμα δεν νομίζω ότι αυτή θα ήταν βιώσιμη λύση αν απλώς μειώσουμε τις τιμές. Ε, επειδή υπάρχει μια τεχνική λύση, ο κύριος Κρόιτσμαν αναφέρθηκε ήδη και στην ε, δυνατότητα χρήσης τοπικού δικτύου για τις υπηρεσίες δεδομένων, θα πρέπει να καθορίσουμε τα κριτήρια για τεχνικές λύσεις κατά τρόπον ώστε οι λύσεις αυτές να μην αποκλείονται. Ε, ίσα ίσα θα πρέπει να ενθαρρύνονται. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κατά πόσον είναι αποτελεσματικές ως προς το κόστος οι διάφορες τεχνικές λύσεις. Αλλά αυτή είναι μια πολύ σημαντική τεχνική ε, πτυχή την οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Όσον αφορά τώρα τα κενά. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που ούτως ή άλλως είπα επανειλημμένος ενώπιον αυτής της Επιτροπής, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Εάν πράγματι θέλουμε να λειτουργήσουν τα διαφορετικά μέσα, αν θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό στην αγορά, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε να υπάρχουν και νέοι παράγοντες στην αγορά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μεταπόληση ε, ή και νέους παράγοντες, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και νέους παρόχων. Άκουσα μία ή δύο φορές τις λέξεις ολιγοπόλιο και μονοπόλιο εδώ. Ε, η συμπεριφορά της αγοράς, αν θέλουμε να αλλάξει, θα πρέπει να δημιουργήσουμε αλλαγή και να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω των κατάλληλων διαφορετικών μέτρων. Δεν θα ήθελα και πάλι να λάβω θέση ε, για το επίπεδο των ανωτάτων ορίων, αλλά νομίζω ότι άκουσα αρκετές παρατηρήσεις που έλεγαν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε τουλάχιστον με τα κοινά σε θέματα χονδρικής πώληση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταγωνιστών στην είσοδό του στην αγορά. Η πρότασή μας βασίστηκε στις εκτιμήσεις κόστους Μπάραξ, αλλά ε, νομίζω ότι ο τομέας της χονδρικής πώληση είναι το κλειδί αν θέλουμε να ενισχύσουμε την εισαγωγή στην αγορά και να άλλων παρόχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Τζιμ Νίμπλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για δύο λεπτά όπως μου ζητήσατε. Δύο λόγια για τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι επικεντρώνονται στον ανταγωνισμό από ό,τι άκουσα σήμερα εδώ στην αίθουσα αλλά και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και από τις εκθέσεις του Συμβουλίου στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εισαγωγή διαρθρωτικών ε, μέτρων για να υπάρχει η λεγόμενη δυνατότητα αποσύνδεσης ώστε ο κάθε ε, καταναλωτής μπορεί να επιλέξει περιαγωγή από τον ε, πάροχό του. Υπάρχει και κάτι όμως το οποίο δεν δίνεται ιδέουσα προσοχή, είναι η ανταγωνιστική αγορά για τα τοπικά πακέτα περιαγωγής και εδώ είναι ο πραγματικό στόχο αυτού του κανονισμού να έχουμε τιμές περιαγωγέ παραγωγής που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ε, τιμές ε, ε, στη χώρα του καθενός. Ο ανταγωνισμός τώρα για τα πακέτα είναι αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα είναι αυτό το οποίο θα επιλέγουν οι περισσότεροι καταναλωτές. Προτιμούν να έχουν μία λύση και όχι να έχουν ένα μείγμα από διάφορους παρόχους. Ε, θέλουμε να έχουμε λοιπόν χονδρικές τιμές οι οποίες θα είναι πολύ πιο κοντά στο ε, κόστος στο εσωτερικό της χώρας του καθενός. Ε, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ε, δεν μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή απευθείας, ε, δεν μπορούμε να έχουμε κόστος που να είναι χαμηλότερο από το εσωτερικό κόστος, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Οι προτάσεις του κυρίου Άγκστρομ όσον αφορά τα data για παράδειγμα να υπάρχει μια τιμή χονδρικής ε, ε, με ανώτατο όριο στα 10 ευρώ ανά gigabyte αν οι τιμές χονδρικής φτάσουν σε αυτό το επίπεδο τότε σίγουρα θα διευκολύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα μπορούν να παρέχουν ένα πακέτο εσωτερικών ε, υπηρεσιών και παρουσιών περιαγωγής σε ανταγωνιστική τιμή. Κάτι το οποίο επιπλέον θα επιτύχουμε θα είναι να μην εισέλθουν στην αγορά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία είσοδος μέσω αποσύνδεσης ε, της ε, τιμής ε, εάν θέσουμε το ανώτατο όριο της λιανικής πώλησης στα 20 ευρώ ανά γιγαμπάιτ. διότι δεν θα υπάρχουν ε, δυνατότητες για νέες ε, ε, δουλειές σε τέτοιο επίπεδο. Εξαρτάται λοιπόν τι ανταγωνισμό θέλετε να ευνοήσετε. Θέλετε ανταγωνισμό μεταξύ πακέτων εσωτερικών και υπηρεσιών και υπηρεσιών παραγωγής ή θέλετε να έχει έναν ανταγωνισμό όπου οι πελάτες θα επιλέγουν διαφορετικό πάροχο από τον πάροχο που έχουν στη χώρα τους. Κάποιοι θα επιλέξουν τη μία λύση, άλλοι την άλλη. Θα πρέπει να βρούμε μία κατάλληλη ισορροπημένη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση ως προς τις επιλογές και όχι ενίσχυση των υπαρχουσών δομών της αγοράς, κάτι το οποίο δεν είναι σοφό για την, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Και η κυρία Κόρχολα τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολιτικό χριστουγεννιάτικο δώρο. Ε, βεβαίως είναι πολιτικό όνειρο το να ασχοληθεί κανείς και να ζητήσει λύση για ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να διορθωθούν για να κάνουν τη διαφορά υπέρ του καταναλωτή. Και τώρα για λίγο θα κάνω χρήση της μητρικής μου γλώσσας. Ο στόχος λοιπόν είναι σε κάποια φάση να μην χρειάζεται πλέον ρύθμιση να μην υπάρχουν κανονισμοί. Ε, ε, παρόλο που θα υπάρχουν διαφορές στις τιμές. Ε, κύριε Λαβέλα, πράγματι είναι λογικό αυτό που λέτε. Στον κύριο Κρότσμαν λέω ευχαριστώ, είναι σπουδαίο που κατανοήσατε την ουσία της έκθεσής μου. Είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή να διασφαλιστεί η ύπαρξη του ανταγωνισμού και να ε, προληφθούν ολιγοπολιακές καταστάσεις. Γι' αυτό η αναζήτηση μιας ισορροπίας είναι απαραίτητη. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, και αναφέρομαι και σε άλλες επιτροπές, σε πολλές συζητήσεις αναφέρθηκε ε, αναφέρθηκαν ε, εθνικές προσφορές τιμών ή εθνικός καθορισμός, ε, καθορισμός τιμών σε εθνικό επίπεδο. Τιμές μάλιστα οι οποίες θα είναι βιώσιμες στο εξωτερικό. Ελπίζω ότι το επίπεδο αυτό θα είναι παρόμοιο, παρεμφερές, αλλά αυτή η, η υπερβολικά καλή τιμή δεν είναι ενδεικτική ε, του πραγματικού κόστους, διότι το τρέχον έσοδο από την περιαγωγή είναι πάρα πολύ υψηλό. Τα έσοδα από την περιαγωγή ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να επιδοτηθούν προσφορές στην λιανική. Ε, ελάχιστοι χρήστες ε, έξυπνων τηλεφώνων αγοράζουν φθηνά gigabytes. Ελάχιστοι άνθρωποι χρειάζονται αυτούς τους όγκους. Άρα λοιπόν οι προσφορές είναι υπερμεγέθης αλλά άχρηστες. Χίλια μεγαμπάιτ ας πούμε αγοράζει κανείς. Να τα κάνει τι όμως. Ένας 300 μεγαμπάιτ χρησιμοποιεί ένας συνηθισμένος χρήστης του iPhone. Άρα λοιπόν μιλούμε για μεγάλους όγκους σε αυτή την περίπτωση που είναι κατανοητό όταν πολύ κανείς ένα πακέτο αλλά δημιουργεί μία εντύπωση ε, χωρίς ε, λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θαυμάσια συζήτηση και σας εύχομαι όλους καλά Χριστούγεννα. Ο Πρόεδρος, θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε τώρα το χρονοδιάγραμμα και έχω και μία ακόμα ανακοίνωση να κάνω πριν φύγουμε. Άρα λοιπόν, προθεσμία τροπολογιών αύριο στις 12. Θα τις εξετάσουμε στις 6 Φεβρουαρίου και σχεδιάζουμε να ψηφίσουμε την ίδια μέρα προς το παρόν, διότι και η Επιτροπή Βιομηχανίας θα ψηφίσει στις 22. Θα επιταχύνουμε λοιπόν τη διαδικασία στο, μέγιστο, στο πλαίσιο του δυνατού και ελπίζω να υπάρχει επαρκής χρόνος για να συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα πάει στην Ολομέλεια στα μέσα Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και τέλος θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι εξ ονόματος του εισηγητή Εύγιου Κόσνεστικ που έπρεπε να επιστρέψει στην Τσεχία επειδή έπρεπε να παραστεί στην κηδεία του πρώην Προέδρου Βάσλαβ Χάβελ κυκλοφόρησε ένα πρόγραμμα που δείχνει το τελικό αποτέλεσμα της Συμφωνίας του Προϋπολογισμού. Και θα δείτε εκεί το τι ακριβώς προτείνει αυτή η Επιτροπή. Σε γενικές γραμμές ε, κερδίσαμε σε κάποια, χάσαμε σε άλλα, αλλά πάντως η πρόταση είναι ελαφρώς αρνητική, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι μια αποδεκτή λύση. Υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με κονδύλια σε κάποια κεφάλαια αλλά νομίζω ότι ο κύριος Κόσνιτσικ έκανε πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν η Σκιώδης ε, η θα ήθελε να προσθέσει. Όχι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, τους διερμηνείς που μας έδωσαν πρόσθετο χρόνο και τώρα με μεγάλη χαρά θα κλείσω αυτή τη συνεδρίαση θα ευχαριστήσω τον Ρόνταν για όλα όσα έκανε ως επικεφαλής ε, αυτού του τμήματος. Εγώ ήμουν ένας από τους τρεις προέδρους που προείδρευσαν στην Επιτροπή αυτή και η προηγούμενη ήταν ο Άλλη Μακάρθη και ο κύριος Ε, δουλέψαμε λοιπόν πολύ ε, και συνεργαστήκαμε μαζί του. Έχουμε τώρα ένα μικρό κοκτέιλ κατάλληλο για την εποχή και με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε και όσους διερμηνείς θα ήθελαν να παραστούν σε αυτήν την μικρή δεξίωση. Πέραν αυτών θα ήθελα να σας ευχηθώ πολύ καλά Χριστούγεννα, χαρούμενη νέα χρονιά και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και με χαρά θα σας ξαναδώ τον Ιανουάριο.